Καλημέρα, Επίτροπε Γκάμπριελ. Καλημέρα, συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. The uh, Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις παρατηρήσει, θεωρείται εγκριθή σε ημερήσια διάταξη. Και ε, αν δεν υπάρξει επομένω κάποια... Α, ναι, συγγνώμη, ε, ε, εκτός από το σημείο υπαριθμών 5, θα μεταδίδεται στο ίντερνετ η συνεδρίαση όλη. Στις 11 η ώρα θα αρχίσουμε αυτή την μετάδοση. Με αυτό το δίκτυο mainstreaming. Ε, ανακοινώσεις της Προέδρου ε, έχουμε τις ιδέες της 27 Σενάτου και οπότε και αποφάσισαν οι συντονιστές να υιοθετήσουν κάποια τοποθέτηση υπό την μορφή ε, τροποποιήσεων και τροπολογιών για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία όσον αφορά το ΕΛΚ και έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις για την απαλλαγή ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό 2019 όπου είναι η συγκεντρική κυρία Μπιόρκ και θα ζητήσουμε την άδεια για κάποιες ε, ακροάσεις στην περίοδο Νοέμβριος με τέλος της θητείας όσον αφορά την ε, προσχώρηση στη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης για μελέτες Ουγγαρίας και κάποιες άλλες εκδηλώσεις εν των εκλογών και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για τη βία κατά γυναικών και τον ρόλο της ε, γυναίκας στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Έχουμε τις εξής αποστολές. Γερμανία και Ισπανία. Είπαμε για την πολέμηση της ε, βίας και για τον ρόλο της ε, γυναίκας σε ειρηνευτικές διαδικασίες. Αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Προχωρούμε στη μέση. Διάταξε το πρώτο σημείο είναι η επίσκεψη της της Μαρίας Γκαμπριέλ της ε, Επιτρόπου για Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή ε, Γενικών Υποθέσεων στις 9 ε, η ώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση των Επιτρόπων και ευχαριστούμε όμως που εσείς ήρθατε. Ευχαριστούμε που βρήκατε λίγο χρόνο τόσο ώστε να έρθετε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση. Για τα δικαιώματα των γυναικών σε σχέση με το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Έχετε την σκητάλη εσείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές και βουλευτίνες της Επιτροπής ε, γυναικών. Ευχαριστούμε που με καλέσατε και να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να έρχομαι εδώ. Γνωρίζω την Επιτροπή επί σειράν ετών ήμουν Ευρωβουλευτής. Έχω μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά σας, γιατί πολλές φορές φέρουμε κάποια πράγματα η αυτονόητα, κάποια πράγματα συνέχεια είναι στην επικαιρότητα, μα είναι ζητήματα που καίνε την κοινωνία, ε, έχουν σχέση με ε, δημοκρατικές αρχές ε, και βασικά μας πιστεύω, οπότε να δούμε κάποιες σκέψεις, να δούμε κάποιες δράσεις που αναλάβαμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια της ψηφιοποίησης να αναβαθμιστεί η γυναίκα όταν έλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο, το πρώτο μου ερώτημα ήταν έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική για τις γυναίκες. Η απάντηση ήταν αρνητική και κινητοποιήθηκε το επιτελείο μας και μέσα σε πέντε μήνες επεξεργαστήκαμε τέτοια στρατηγική που είναι μια αφετηρία. Από το 2013 για πρώτη φορά κάναμε μια μελέτη σύμφωνα με αυτήν έχουμε κάποια στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφιακά έχει τάση αρνητική. Και από πολλές πλευρές αυτό. Όταν ε, αναφερόμαστε σε αυτούς που δουλεύουν με ψηφιακή τεχνολογία, από 8 εκατομμύρια ειδικού μόνο 17% είναι γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. είχαμε 350.000 ειδικέ και το 2020 θα είναι 500.000. Μα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την κοινωνία και για την οικονομία. Επομένως θα δούμε θα, πώς θα μπορέσουμε να ε, αναβαθμίσουμε τις γυναίκες που θα ωφελήσει κατά 16 δις. Οπότε αν εξετάσει κανείς τι ισχύει όσον αφορά τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες για αυτούς τους κλάδους και ε, σε κάθε 100 αποφύντους από αυτές τις σπουδές είναι 24 γυναίκες και μόνο 6 κάνουν μια σταδιοδρομία. Ενδιαφέρονται τα κορίτσια για την τεχνολογία τώρα πια και θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο σε αυτούς τους κλάδους και μετά στην αγορά. Και όταν μιλούμε για την επιχειρηματικότητα έχουμε μόνο 17% γυναίκες που είναι σε αυτούς τους κλάδους επιχειρηματίες. Και βλέπουμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις των γυναικών έχουν 3% ε, θετικά αποτελέσματα χρήση σε σχέση με επιχειρήσεις ανδρών. Οπότε έχουμε μία στρατηγική με τρεις άξονες. Πρώτα πρώτα να συνεχίσουμε την καταβλέψη των στερεοτύπων. Είναι σαφές ότι σήμερα οι νέες γυναίκες χρειάζονται έμπνευση, χρειάζονται την αυτοπεποίθηση, role models χρειάζονται, πρότυπα. Όλοι που κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Δεύτερος άξονας αφορά το πώς θα ελκύσουμε περισσότερες νέες γυναίκες σε αυτούς τους κλάδους της ε, παιδείας που αναφέραμε. Οπότε έχουμε και μια σειρά σχετικών πρωτοβουλειών. Να, να σας πω μία που έχει συμβολική σημασία. Ξεκίνησε στις 6 Δεκάτου, θα συνεχιστεί μέχρι τις 21 Δεκάτου. Είναι αυτή που ονομάζεται European Code Week και έχουμε ένα σωρό εθελοντές οι οποίοι ε, προτάσουν το ότι έχουμε την καινοτομία, δεν πρόκειται ποτέ να μας αντικαστήσουν τα ρομπότ, ούτε η τεχνολογία. Για πέρσι, αυτή η εβδομάδα, είχε πάνω από ένα εκατομμύριο 200.000 ε, συμμέτοχους, ούτως είπε 46% ήταν γυναίκες και τον Απρίλιο απίθυνα επιστολή προ όλους του υπουργού παιδεία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και του είπα ότι θα πρέπει να προαγάγουν την συμμετοχή των νέων γυναικών. Και τους κάλεσα να συμβάλλουν σε αυτές μας τις φιλοδοξίες και να καλυφθούν 50% των ευρωπαϊκών σχολείων από αυτή την πρωτοβουλία μέχρι το 2020. Επίσης, είπαμε να προβάλλουμε περισσότερο κάποια έργα, προγράμματα που ενθαρρύνουν τα κορίτσια να συμμετάσχουν. Ας πούμε, έχουμε τα σχετικά βραβεία στα ψηφιακά που θα απονεμηθεί στην Βιέννη το Δεκέμβριο. Για πρώτη φορά έχουμε ένα βραβείο για κάποια project που αφορούν ε, τις νέες γυναίκες. Για δεύτερη φορά θα γίνει αυτή η εκδήλωση και θα κινητοποιηθούμε ούτως ώστε όλη αυτή η υπόθεση να αποκτήσει περισσότερη προβολή. Επίσης ο τρίτος άξονας αφορά την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συμβάλλουμε σε κάποια project τα οποία να προβάλλουν αυτή την πλευρά των γυναικείων δραστηριοτήτων, να ενθαρρύνουμε τις νέες γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες και μόλις μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο να μπορέσουν να εξελιχθούν, να ανέβουν. Οι αναλύσεις λένε ότι και εδώ υπάρχει χάσμα, πρόβλημα. Οπότε τον ε, Ιούνιο έχουμε μία διάσκεψη Digital for Her. Οπότε θα έχουμε διάφορο από τον δυτικό κλάδο, από μεγάλες εταιρείες, από χρηματοοικονομικά, τηλεπικοινωνίες και όχι μόνο, οπότε θα καταλήξει αυτή η εκδήλωση σε κάποια διακήρυξη και οι εταιρείε θα δεσμεύονται και να έχουν περισσότερες γυναίκες, να έχουν κάποια προγράμματα στα οποία θα καθοδηγούν, θα προπονούν το ΣΥΠΗΝ τις γυναίκες για αυτές τις υποθέσεις. Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδρομή. Έμαθα όταν ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο ότι το, το θέμα δεν είναι στρατηγικές, ε, η θεωρίες, είναι η υλοποίηση και η συνέχεια που δίνεται. Οπότε ε, διαπιστώνουμε ότι η κρίσιμη μάζα είναι πολύ σημαντική και έτσι βγαίνουν αποτελέσματα. Οπότε, με όργανα, ε, σε σχέση με την ισότητα των φύλων, φτιάχνουμε μια πλατφόρμα ούτω ώστε να προβάλλουμε τις εταιρείε που κάνουν πράγματα για τις γυναίκες. Άριστες πρακτικές, τις προβάλλουμε, ε, τα προγράμματα, τα αξιόλογα και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και οπότε έτσι ελπίζουμε να κάνουμε βήματα πρώτο σύντομα για να δούμε και κάτι άλλο το οποίο ξέρω ότι σας ενδιαφέρει γιατί και το Κοινοβούλιο έχει μια γνωμοδότηση. Κυρία Σόιντροβα, όσον αφορά τον ρόλο των ΜΜΕ όταν μιλούμε για καταπολέμηση στερεοτύπων, ε, λέμε ότι θέλουμε να ελκύσουν περισσότερες γυναίκες, να προβάλλουμε την επιχειρηματικότητά τους. Ε, άρα τα ΜΜΕ είναι πολύ σημαντικά και τον ε, Μάρτιο που είχαμε στην Κροατία κάποια σύνοδο έλεγα ότι εκεί πρέπει να δούμε τι λέει η νομοθεσία, ποιοι είναι οι φραγμοί, ποιες είναι οι πρακτικές και ζήτησαμε να γίνει μια έκθεση. Ε, αυτή είναι έτοιμη τώρα το Σεπτέμβριο να την μελετήσετε γιατί έχει αξιόλογα συμπεράσματα. Όχι μόνο υπάρχει η υποεκπροσώπηση, αλλά φύγονται οι γυναίκες και από τα στερεότυπα σε κράτη-μέλη όπου ξεκάθαρα οι γυναίκες, μόλις εμφανίζονται στην ε, τηλεόραση, έχουν δύο ρόλους. Ή είναι super models ή είναι καλές νοικοκυρές. Ε, βέβαια, και αυτό δεν είναι συγκερασμός επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Στην έκθεση εκείνη, ξεκάθαρα αναδεικνύεται ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε εκπομπές σοβαρές εντός εισαγωγικών ως ειδικοί, ως εμπειρογνώμονες. No Women No Panel. Μια τέτοια εκστρατεία ξεκίνησα και είπα ότι δεν πάω σε κάποια εκδήλωση όπου είμαι η μόνη ομιλήτρια, όπου δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Πιστέψτε με. Αυτό έπιασε. Απέδωσε αποτελέσματα. Έχουμε τώρα παραδείγματα. Το πήραν το μήνυμα οι οργανώτες. και σε κάποια εκδήλωση άλλαξε το πρόγραμμα και μας ειδοποίησαν σχετικά. Να, πώς θα μπορέσουμε κάποιες γυναίκες με ειδικές γνώσεις να τις προβάλλουμε. Δεν, δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν το σκέφτονται, δεν τους ενδιαφέρει τους οργανωτές. Ε, να, επομένως ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Επίσης, άλλη πρωτοβουλία σε υπουργικό επίπεδο το Σεπτέμβριο με την Αυστριακή Υπουργό οργανώσαμε ένα πρόγευμα. Και είπαμε ότι θέλουμε αυτά τα θέματα να ανέβουν σε υπουργικό επίπεδο και ότι θέλουμε σε τακτά διαστήματα αυτά να απασχολούν τις ε, ομάδες εργασίας ε, ψηλού επίπεδου και εισηγηθήκαμε αυτά τα οποία σας έχει στείλει η γραμματεία. Και στην έκθεση του Μαΐου όλα αυτά θα τα περιλάβουμε, τα στοιχεία αναχώρα για την συμμετοχή των γυναικών στα ψηφιακά. Και στις δικές σας φαντάζομαι υπάρχουν κάποια στερεότυπα ε, αλλά αν κάνουμε μια ξεκάθαρη καταγραφή της κατάστασης κάθε χρόνο, ε, τότε μπορούμε να εστιαστούμε στις άριστες πρακτικές και έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι για την κατάσταση, για την πρόκληση αυτή. Να μην με γρηγορήσω, αλλά ήθελα να σας πω τι κάναμε αυτή τη χρονιά. Έχουμε αυτή τη στρατηγική, τους τρεις ε, άξονες, τον Ιούνιο, πρόγραμμα δράσης, συγκεκριμένα παραδείγματα. Και σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει η κινητοποίηση να συνεχιστεί. Ε, τα ψηφιακά είναι κάτι που εξελίσσονται κάθε μέρα. Δεν θα πρέπει κανείς να χάσει το τρένο. Θα πρέπει οι γυναίκες να μπορέσουν να δουλεύουν ε, με αυτοπεποίθηση και να αξιοποιείται το ταλέντο τους, η ικανότητα τους υπέρ όλων, υπέρ της οικονομίας, υπέρ της κοινωνίας. Αυτά και ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε για την παρουσίαση αυτή και θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Αγνέσσα Κοβλώστα έχει πρώτα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι σας θαυμάζω και θαυμάζω τα όσα έχετε καταφέρει. Νομίζω πως είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι είστε επίτροπος και έχετε φτάσει ε, σε μια τόσο υψηλοβαθμή θέση γιατί είναι λίγοι οι οποίοι κατέχουν μια τέτοια θέση και οι οποίοι αναφέρονται τόσο συχνά στα ζητήματα τη διάσταση του φύλου. Πρόκειται δηλαδή για μια πάρα πολύ καλή πρακτική την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις στρατηγικές και τα σχέδια δράση που έχετε προτείνει. Και θα ήθελα επίση να θέσω ένα ερώτημα. Παρά όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε και όλε αυτέ τι ιδέε οι οποίες έχουν προωθηθεί υπάρχουν ακόμα που πολλά ε, υπάρχουν ακόμα πολλά που θα πρέπει να κάνουμε και νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ από το επίπεδο της ε, παιδείας. Γιατί τα προβλήματα αρχίζουν να ε, διαφαίνονται στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Ε, οπότε, ε, παρότι πρόκειται βέβαια για ένα ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, υπάρχει εδώ ο τομέας ε, της παιδείας ε, ε, στο πλαίσιο του οποίου συνέρχονται οι Υπουργοί Παιδείας και μάλιστα και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση εκεί. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν ευκολότερα να περνούν αυτό το χάσμα το ψηφιακό εάν το σύνολο της εκπαίδευσης γινόταν πιο ψηφιακό. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα η ηλεκτρονική μάθηση διαποστάσεω δηλαδή, εμ, γινόταν ευκολότερη, γιατί κάτι τέτοιο θα απέβαινε προ όφελο ε, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Έριξα ε, μια ματιά στο έγγραφο το, το δικό σα και διαπιστώνω ότι ακόμα και στην Εστονία, όπου δηλαδή υπάρχει υψηλό βαθμό ψηφιοποίηση, ε, παραμένουν οι ίδιε διαφορέ σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε και γενικότερα την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα και επιχαίρω το γεγονός ότι εργάζεστε από αυτό. Ε, καθώς βέβαια το, ε, μέσα με το μερίδιο της ε, ψηφιακής οικονομίας ε, έχει αρχίσει να μειώνεται αντί να αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρος η κυρία Μαρία Νόγκλα έχει το λόγο. Ε, Σα είδα σήμερα εδώ το πρωί και θυμήθηκα και την αποστολή στην οποία είχαμε βρεθεί από κοινού στην να Φάσο. Χαίρομαι λοιπόν που σα βλέπω ε, εδώ σήμερα και ε, μου αρέσει το γεγονό ότι αναφέρεστε με προοδευτικό τρόπο στα δικαιώματα των γυναικών. Ήταν πραγματικά μια προοδευτική παρέμβαση την οποία κάνατε και η οποία θα μπορούσε να έχει προέλθει από την δική μου παράταξη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή. Αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν κατάφερε να προωθήσει την ε, υιοθέτηση μια στρατηγική σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Και τώρα μας αναφέρεται ε, πως ε, προβλέπεται μια ε, στρατηγική σε τρει επιλώνε σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να σα ε, ε, καλέσω να μιλήσετε μια ακόμα φορά με τον πρόεδρο Γιούκερ και με τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπή ω προ το πώ ήταν δυνατόν στο πλαίσιο αυτή τη Επιτροπή και με εσέ ω Επίτροπο να μην καταφέρει η Επιτροπή να επιβάλλει μια τέτοια στρατηγική σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων. το ότι δηλαδή οι ε, διάφορες σκέψεις τις οποίες είχαμε κάνει για παράδειγμα από το 2014 ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα έγγραφο εργασίας απλώς και μόνο και όχι ένα έγγραφο στρατηγικής. Δηλαδή από τότε ξεκίνησε μια χώρισε εδώ σε σχέση με αυτό το ζήτημα και ε, επειδή στη δική σα παρέμβαση αναφέρεστε σε μια στρατηγική ε, με τρει πυλώνε, με σαφήνεια, θα ήθελα να σα πω ότι δεν χρειαζόμαστε μια στρατηγική ε, τέτοιου είδου μόνο στον τομέα της, ε, ε των ψηφιακών τεχνολογιών και τη ε, πληροφορικής, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τη ισότητα των φύλων και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μιλήσετε με τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ για αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την εξάλληψη των ε, στερεοτύπων, γνωρίζετε πω με την αύξηση της ε, δεξιάς η ο ρόλος της γυναίκας παραπέμπεται και πάλι στην, ε, ε, στην, ε, στον οίκο, στα του οίκου και στα παιδιά. Και νομίζω πως αυτή η οπισθοχώρηση και εδώ η οποία δείχνει να εμφανίζεται παντού, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ακριβώς Αναφέροντα το επιχείρημα ότι οι γυναίκε δεν είναι απλώ και μόνο μητέρε. Βλέπουμε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Πολωνία που γίνεται μόνο λόγο γίνεται λόγος ξανά ξανά και αναφέρονται μόνο στις, ε, στις ε, γυναίκες ως ε, μητέρες. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη προσπάθεια και να μην ξεχνάμε δηλαδή όλα τα άλλα ζητήματα και να μην εστιάζουμε μόνο στην ψηφιοποίηση. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών. Γιατί ακόμα κάποιοι δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί υπάρχουν ε, κάποια έγγραφα τα οποία κυκλοφορούν σήμερα ημέρα τα οποία αναφέρουν πόσα παιδιά θα πρέπει να έχει μια γυναίκα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανταπαραγωγικά, δεν μα βοηθάνε. Οπότε αυτό που σα καλώ να κάνετε, κυρία Επίτροπε, είναι να έχετε πάντα κατά νου την συνολική εικόνα. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία. Νίμπλερ, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, εισηγήτρια. Να σας συγχαρώ για τη στρατηγική την οποία υποβάλλατε και για το γεγονός ότι συμπεριλάβατε το θέμα αυτό στις προτεραιότητές σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό ότι ε, κοιτάξατε τα γεγονότα και έγινε ανάλυση σχετική σε, σε επίπεδο κρατών μελών. Και αυτό κατέδειξε πόσο δραματική είναι η κατάσταση σε τελική ανάλυση και πόσες... Ε, ευκαιρίες μπορεί να έχει η, η ψηφιοποίηση και πόσο αμελείται στην παρούσα φάση. Στη στρατηγική σας λοιπόν ε, τα διάφορα στοιχεία τα οποία μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνος. Θα ήθελα να δείξω μόνο δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία όλου ο ιδιωτέρως γιατί και εγώ στο Μόναχο στην περιοχή μου διοργάνωσα μια ημερίδα ένα συνέδριο επί δύο ημέρες ε, για το θέμα της ψηφιοποίησης και είχαμε λοιπόν πολλούς εμπειρογνώμονες και τους βάλαμε στο έτρανο και τους ρωτήσαμε γιατί τα κάνετε αυτό ως τώρα. Γιατί λοιπόν στραφήκατε πιο στην ψηφιοποίηση και η, το, η απάντηση, το αποτέλεσμα ήταν ότι είναι απογοητευμένες πολλοί οι γυναίκες ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Χτυπούν ε, σε αδιέξοδο και γι' αυτό λοιπόν στρέφονται στην ε, ψηφιοποίηση και σε ό,τι αφορά την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Απέραντες είναι οι ευκαιρίες για τις γυναίκες να αναξαρτοποιηθούν, να κάνουν να, ανοίξουν επιχειρήσεις ε, ανεξάρτητα από άλλους Αυτές οι αλλαγές λοιπόν που επιφέρει η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να φοβίζουν πολλούς. Αλλά θέλουμε να τη και να δώσουμε μορφή στην ε, κοινωνική αυτή εξέλιξη και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει για την κοινωνική αποδοχή των εξέλιξεων αυτών. Και εδώ έχει σημασία το πρόγραμμα πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις τομές ε, στην ε, εξέλιξη. Πώς θα φροντίσουμε λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή για τα μέσα αυτά, για την παγκοσμιοποίηση την ίδια, για τις προκλήσεις της ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να δώσουμε πιο πολλά επιστημονικά τεκμήρια. Άλλα δύο σημεία να αναφέρω. Το θέμα της, ε, του πρασινίσματος των επιχειρήσεων και εδώ θα ήθελα να πω ότι υπέβαλε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ευκολύνει αυτό σε περίπτωση αποτυχίας να υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία, μια αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Και εδώ πέρα λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει το στίγμα του. Ξεκινάνε οι τριμερείς διάλογοι, αλλά σημειώνω ότι πολλές γυναίκες ανησυχούν ότι αν πάρουν ένα ρίσκο και δημιουργήσουν μια επιχείρηση και δεν πετύχουν με την πρώτη, τι συμβαίνει. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει αυτό το στίγμα της αποτυχίας. Ενώ στην Αμερική, στην Αμερική υπάρχει η αντίληψη πιο πολύ ότι ακόμα και αν κάποιος έχει σημειώσει πολλές αποτυχίες, αυτό μετράει ως εμπειρία. Άρα, να υπάρχει αυτή η δεύτερη ευκαιρία ακόμα και σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας. σημαντικό. Τελευταίο στοιχείο No Women, No Panel. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρώ είναι εξαιρετική. Θα την προωθήσω και στο πολιτικό μου κόμμα. Δεν είναι δεδομένο ότι εκπροσωπούνται οι γυναίκες όπως πρέπει σε μεγάλα πάνελ και επιτροπέ. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε και φυσικά είναι πολύ σημαντικά και τα μέσα ενημέρωση εδώ. Οι εκπομπέ που προβάλλονται ε, πιο πολύ στη Γερμανία είναι η Heidi Klum, το επόμενο top model της Γερμανίας. Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Αυτά τα στερεότυπα ακόμα επικρατούν σε ό,τι αφορά τα δημόσια πρόσωπα. Οι καταλαβαίνετε, είναι κατανθουσιασμένοι. Όπου μπορούμε όμως και όπου έχουμε την ευκαιρία κάτι να φροντίσουμε να αλλάξει αυτό το πρότυπο και σε ό,τι αφορά λοιπόν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ψηφιοποίηση. Και νομίζω ότι το βασικό είναι να προβάλλουμε τα σωστά παραδείγματα ξανά και ξανά και ξανά σε εφημερίδες, τηλεοράσεις και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ. Και να με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Αλλά το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα που περάσαμε ακούσαμε το θέμα της ψηφιακής, ε, του ψηφιακού προγράμματος και με είχε συναρπάσει. Ε, να ξεκινήσω με την πρωτοβουλία No Women, No Panel. Μία από τις πιο καλές ε, πρωτοβουλίες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντική. 51% του κόσμου είναι γυναίκες. Πώς να το κάνουμε, θα πρέπει να εκπροσωπούμαστε σε κάθε πάνελ. Υποστηρίζω την ε, πρωτοβουλία αυτή. Να σας συγχαρώ και προσωπικά, κυρία Γκάμπριελ, γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο καταφέρατε να τα προωθήσετε όλα αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει το θέμα της ισότητας των φύλων, το θέμα της διάστασης του φύλου και στην ψηφιοποίηση και αυτό να προσεγγίσει τους πολίτες. Είναι εξαιρετική αυτή η στρατηγική και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την οικονομία μας. Καλωσορίζω λοιπόν την πρωτοβουλία σας και πραγματικά πρόκειται για μια πολύ καλή αρχή. Υπάρχουν όμως διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως ξέρετε κάποιοι διατείνονται τα, τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με κούκλες γιατί αυτό επιτάσσουν τα γονίδια τους ενώ τα αγόρια αντίστοιχα μπορούν να παίζουν με αυτοκινητάκια. Δεν ε, πιστεύω σε αυτά τα στερεότυπα. Θεωρώ ότι το παιδί είναι ελεύθερο για όλους. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε λοιπόν τα συστήματα εκπαίδευσή μας και πιστεύω ότι εκεί υστερούμε στην παρούσα φάση. Η κυρία Γκάμπριελ και η υπόλοιπη επιτροπή. Θεωρώ ότι κάνουν καλή δουλειά. Συνεχίστε λοιπόν. Σας υποστηρίζουμε απόλυτα. Ευχαριστούμε την κυρία Ντουμπράφκα Σουίτσα και τώρα να δώσω το λόγο πάλι στην Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας γιατί θεωρώ ότι αυτό που μας δίνουν οι παρεμβάσεις σας είναι η υποστήριξη. Αυτό χρειαζόμαστε και όντως πριν από ένα χρόνο υπήρχε η στρατηγική για τις γυναίκες, για την ψηφιοποίηση. Η απάντηση ήταν όχι και να προσθέσω ότι όταν το ρώτησα αυτό μου απάντησαν ότι μα δεν έχουμε χρόνο κυρία Επίτροπε μέχρι το τέλος της θητείας. Αρνούμε να δεχτώ αυτή την απάντηση. Ακόμα και ένα λεπτό να υπάρχει Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά σε δύο χρόνια, αλλά να έχουμε πρωτοβουλίε και δράσει που θα ενθαρρύνουν τι γυναίκε. Αυτό λοιπόν αρκεί και είναι καλύτερα από το να μην κάνουμε τίποτα και να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξη. Για τι ερωτήσει που μου ετέθησαν, Αγνιέσκα, ναι, πιστεύω ότι η παιδεία και η εκπαίδευση παραμένουν το βασικό θέμα. Με του υπουργού παιδεία λοιπόν και τι επιστολέ που ε, έστειλα Έχω λάβει ως τώρα 18 απαντήσεις. Ε, μου λοιπόν είναι καμία δεκαριά ακόμα λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τους Υπουργούς ε, Παιδείας να καταρτήσουν ένα κατάλογο βέλτιστων πρακτικών που υφίστανται στις χώρες τους σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κοριτσιών στην ψηφιοποίηση και ήθελα λοιπόν να διεξαγάγω μια σχετική ανάλυση και πριν το τέλη του έτους να δώσω ε, ένα κατάλογο, να προβάλλουμε ένα κατάλογο με τις βέλτιστες πρακτικές ε, Εννοείται ότι δεν είναι ίδιος ο βαθμός ε, προσοχή στο θέμα αυτό από όλες τις χώρες. Έχω ζητήσει λοιπόν πρωτοβουλίες από τις χώρες αυτές ε, και κάποιοι έχουν καταρτήσει πρωτοβουλίες, κάποιοι όχι. Σε ό,τι αφορά όμως την παιδεία, την εκπαίδευση, την ψηφιοποίηση, να σας πω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μεγαλύτερη προσοχή όταν κατέφθασα λοιπόν ε, στη θέση μου, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, είχα θέσει ως πρώτη προτεραιότητά μου την ψηφιοποίηση, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε στους πολίτες. Τα στοιχεία, τα αριθμητικά είναι εξαιρετικά ε, ανησυχητικά. 45% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν τέτοιες ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες. Ξέρετε πόσο είναι αυτή σε εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο, ότι μεγάλο ποσοστό των πολιτών δεν χρησιμοποιούν διαδικτύο. Τώρα θα πρέπει να δράσουμε. Τώρα λοιπόν αρχίσει σταδιακά μια συνειδητοποίηση. Χθε ε, παρευρέθηκα σε μια υπουργική συνάντηση στο Ελσίνκι για την τεχνητή νοημοσύνη και είμαι ενθουσιασμένη που διαπιστώνω ότι οι Υπουργοί Οικονομικών αποδέχθηκαν να εξετάσουν το θέμα αυτό και να εξετάσουν όλος ιδιαίτερος την ψηφιακή διάσταση και αυτό θεωρώ ότι θα μας φέρει αντιμετωπίσουμε τα πρώτα εμπόδια. Καταρχάς ένα θέμα είναι ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα πολλών διαφορετικών ε, υπουργών σε επίπεδο ε, κρατών μελών. Ε, υπουργοί πολιτισμού, υπουργοί παιδείας, Άρα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων χαρτοφυλακίων, προκειμένου να υπάρχει μια συντονισμένη προσέγγιση. Εμείς από πλευρά μα. επιστούμε την προσοχή, μας, ε, την προσοχή των ε, κρατών μελών στο εξή. Ε, με τον Επίτροπο Ναύρατζης δημοσιεύσαμε το σχέδιο δράση για την ψηφιακή εκπαίδευση. Ένα σχέδιο δράση για την ψηφιακή εκπαίδευση. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία σε επίπεδο ε, λοιπόν ε, κράτων μελών ε, θα διοργανώσουμε πιο πολλές ενημερωτικές εκστρατείες, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση των ε, κοριτσιών, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί φυσικά ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δώσει πιο πολύ ε, αυτοπεποίθηση στις κοπέλες, στα κορίτσια, για να τις βάλεις στο σωστό δρόμο. Είναι πάρα πολύ κεντρικός ο ρόλος του εκπαιδευτή, λοιπόν. Και εδώ, λοιπόν, απευθύνω έκκληση και σε εσά ε, για το σχέδιο για να στεφτεί με επιτυχία. Υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει τι πρωτοβουλίε και έχουν εισαγάγει ε, αλλαγέ. Να δώσω το παράδειγμα τη Βουλγαρία, τη χώρα μου, όπου ο Υπουργό ε, Παιδεία από το τρέχον σχολικό έτος αποφάσισε να εισαγάγει <clears throat> στην ε, Δευτέρα Δημοτικού στα παιδιά 8 χρονών μαθήματα για συγγραφή κωδικά. Coding. Όλο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι προαγάγει και την ε, τις αρχές μας, ε, τις πεπιθήσεις μας και παράλληλα θα ενθαρρύνει όλο και πιο πολλά κορίτσια να διαπιστώσουν ότι η ψηφιακή αυτή εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο κάνει κάποιος ε, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ε, ερευνητικά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακολουθήσει ως επάγγελμα. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την, την ψηφιακή εκπαίδευση να υπάρχει ε, μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία και Εθνική Συμμαχία. Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε λοιπόν αυτή η διαδικασία. Σε 1,5 χρόνο λοιπόν καταφέραμε να προσφέρουμε τέτοιες εκπαιδεύσεις σε 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίου πολίτε. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα, στο τοπικό επίπεδο, στο περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο έτσι θα σημειώσουμε αποτελέσματα. Στα πλαίσια λοιπόν τη συμμαχία αυτή ε, διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσει, οι οργανώσει ε, ε, πολιτών όλοι επιμένουν να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των κοριτσιών και θέλω να προβληθεί το θέμα αυτό και στη σχετική ευρωπαϊκή εκδήλωση και έχουμε πλέον λοιπόν ε, ένα, μια επιτροπή διαχειριστική σε ό,τι αφορά τη συμμαχία αυτή για την ε, διανομή των βέλτιστων πρακτικών. Να δούμε τι πρακτικέ έχουν σημειώσει επιτυχία και πώς μπορούμε να τις μοιραστούμε αυτές. Και προφανώ θα το παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό. Και κυρία Νόχιλ, Μαρία, και εγώ θυμάμαι με εξαιρετικέ ε, αναμνήσεις στην αποστολή στην Πουρκίνα Φάσο. Θα ήθελα καταρχάς να επιμείνω στο θέμα των στερεοτύπων. Τον ε, ρόλο που διαδραματίζουμε όλοι μας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τον ρόλο και των μέσων ενημέρωσης, το έθιξε και η κυρία Νίμπλερ το θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και γι' αυτό λοιπόν έχουμε το πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης, μια πολύ συγκεκριμένη α, πρωτοβουλία. Και εδώ και πολλά χρόνια το πρόγραμμα αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε αρεστία στον τομέα των ε, ταινιών. Θα ήθελα να ξέρω τι προγράμματα υπάρχουν και έχουν χρηματοδοτηθεί για τις γυναίκες ε, παραγωγούς και αυτή η ανάλυση έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα, πριν από δύο-τρει εβδομάδε, αλλά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ αρνητικά. Θέλουμε λοιπόν και στον τομέα των μέσων ενημέρωση να υπάρχει προώθηση των γυναικών που παράγουν ευρωπαϊκέ ταινίε. Πώ ε, να προχωρήσουν και τα κορίτσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν ε, δεν ε, αλλάξουμε αυτά τα στερεότυπα, αυτά τα κλισέ δεν θα τοποθετηθώ για το θέμα της στρατηγικής, της ευρωπαϊκής στρατηγικής ε. γενικότερα. Εγώ έχω επικεντρωθεί στο θέμα της ψηφιοποίησης. Προφανώς και υποστηρίζω όλες τις ιδέες που προωθούν α, τα θέματα αυτά. Κυρία Νίμπλερ, Αγγέλικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόθεση της επιχειρηματικότητας στα κορίτσια πάρα πολύ σημαντική και το θέμα της αλλαγής νοοτροπίας. Ναι, προφανώς τη είπα. Όταν κάποιος αποτυχάνει, όταν κάποιος πτωχεύει, δεν είναι χαμένος για μια ολόκληρη ζωή. Αντιθέτως, ε, μια, δύο, τρεις αποτυχίες θεωρούνται ως χρήσιμη πολύτιμη εμπειρία ζωής. Αυτό δεν ισχύει εδώ. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και συνεχίζω να τονίζω το εξής, ότι θέλουμε να συμμετέχουν όλο και πιο πολλέ γυναίκε ε, στην πρόθεση τη επιχειρηματικότητα. Δύο πρωταβουλίες. να τονίσω. Θα γίνει μια σύνοδος ε, ευρωπαϊκών ε, νεοσύστατων επιχειρήσεων τον Νοέμβριο. Θα υπάρξει και ένα βραβείο συγκεκριμένα για γυναίκες. Για τις γυναίκες στην Ευρώπη, αλλά έχω υπόψη μου και τις γυναίκες στα α, Βαλκάνια. Και εκεί θέλουμε να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση, γιατί ξέρετε στην Ήπεθρο στις ε, περιοχές που θέλουμε πιο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ο ρόλος της γυναίκας είναι πιο σημαντικός. Και επίσης το θέμα της βίας θα ήθελα να το θίξω Τον ε, hate speech, ε, των ομιλιών που υποκινούν μίσος. Ναι, σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα νέο κύμα βίας και κυρίως στον ψηφιακό χώρο online. Και ξεκίνησε λοιπόν μια πρωτοβουλία, Safe Internet for the EU, μια εκστρατεία την οποία μπορείτε να προωθήσετε όλοι σας. Και έχω ήδη α, βουλευτές από το Ευρωκοινοβούλιο που προωθούν την πρωτοβουλία αυτή. Η ιδέα είναι απλή, να προωθήσουμε τις δραστηριότητες που ως σκοπό έχουν να διευκρινίσουν ότι και online υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχει ένας χώρος ένομης τάξης. Αυτό θέλουμε να προωθήσουμε. Άρα, απευθυνόμαστε σε τρεις ε, ομάδες. Στους νέους, στους εκπαιδευτές και στους ειδικού ε, του κυβερνοχώρου, τους ε, εμπειρογνώμονες. Το Δεκέμβριο, λοιπόν, θέλω να απονείμουμε το βραβείο αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τα φαινόμενα αυτά στο διαδικτύο. Πρόκειται για θέματα ταμπού, ξέρετε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Ήδη είναι περιορισμένο ο αριθμό των γυναικών στην κυβερνοασφάλεια. Και βέβαια ανακύπτουν και νέες μορφές βίας. Ακόμα και μετά την έναρξη της ε, εκστρατείας μου απευθύνθηκαν online νεαρές κοπέλες που αντιμετωπίζουν παρανοχλήσεις μέσω του διαδικτύου από το σχολείο και παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται αυτές οι τάσεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ότι η φήμη ενός ατόμου, ενός παιδιού μπορεί να εξαρτάται από το πόσα like έχει στο facebook. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε όλα αυτά τα θέματα, να συνεχίσουμε τις εκστρατείες αυτές. Έχουν ήδη διοργανωθεί 15.000 σχετικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση γιατί θέλουμε να υπάρχουν πρεσβευτές σε κάθε χώρα, όχι μόνο πολιτικοί, ξέρετε, συγγραφείς, ε, διασημότητες, αθλητές, για να προωθηθεί η ιδέα αυτή. Σε αυτό το σημείο θα βάλω τελεία και ελπίζω να απάντησα με τον τρόπο αυτό στις ερωτήσεις σας. Και για μια φορά ακόμη πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι προκειμένου αυτή η στρατηγική, αυτή η δράση να μην παραμείνει μια συμβολική δράση, μια υπογραφή σε μια συνθήκη να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα και θέλω να εφαρμόσουμε και να δώσουμε το καλό παράδειγμα μέσω της δικής μας δράσης γιατί πρέπει να αποδείξουμε στα κορίτσια ότι έχουν ευκαιρίες και από εμά εξαρτάται να εξαντλήσουμε το δυναμικό της ψηφιοποίησης. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μην ε, υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση του ψηφιακού δυναμικού αν δεν συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία και οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ και την παρουσίασή σας, αλλά και για την προσωπική ενέργεια που επενδύεται στο να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και ε, σας ευχόμαστε πραγματικά να επιτύχετε ε, τα αποτελέσματα που θέλετε. Η Επιτροπή μας υποστηρίζει όλα αυτά τα βήματα που κάνετε, όλες οι στρατηγικές τις οποίες ε, προωθείτε εδώ, γιατί πραγματικά όλοι χρειαζόμαστε στην ψηφιοποίηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπότιτλοι Uh, dear colleagues, now we will start point four agenda. Πέραμε στο σημείο 4 της μέσης διαταξής. Ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης παγκοσμίω. Ε, αυτό αποφασίστηκε από τους συντονιστές, δηλαδή η διοργάνωση αυτής της συζήτησης για τον ρόλο του γυναικών στην πρόληψη της ε, ριζοσπαστικοποίησης ε, παγκοσμίω. Ε, και οι παρεμβάσεις που θα κάνουν οι ομιλητές μας θα μας επιτρέψουν να αντιληφθούμε καλύτερα το πώς λαμβάνει η χώρα η ριζοσπαστικοποίηση και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της γυναίκες. Καταρχήν θα ακούσουμε παρεμβάσεις από δύο ομιλητές οι οποίοι είχαν προσωπική επαφή με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, ενώ η ακαδημαϊκή διάσταση θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε καλύτερα το πώς λαμβάνει η χώρα η βία ριζοσπαστικοποίηση. Και από εκεί και μετά ε, θα υπάρξει και μία ε, συσχέτιση με την εξωτερική διάσταση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαπιστώσουμε το πώς μπορούμε σε επίπεδο εξωτερική πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωσης να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίηση ανά τον κόσμο. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο ε, στους ομιλητές μας, ξεκινώντα με την κυρία Ντούνια Μπουζάρ, που είναι Γενική Διευθύντρια του CPDSC. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπουζάρ. Πρώτα πρώτα να σας ε, εξηγήσω ε, για τη θέση μου. Το 2014 η κυβέρνηση της Γαλλίας μου ζήτησε να σταματήσω τη δουλειά μου ως ερευνήτρια για να οργανώσω ε, έναν φορέα για τους χίλιους Γάλλους τζιχαντιστές που είχαν γίνει γνωστοί στην αστυνομία είχαν γίνει από Ιράκ και Συρία μέσω της πράσινης γραμμής. Υπήρχε... Ε, ε, δεν ήταν όλοι, ήταν όσες οικογένειες είχαν επισημάνει στην αστυνομία ότι έχουν τζιχαντιστεί δικό τους μέσω της πράσινης γραμμής λοιπόν, από Ιράκ και Συρία. Ήταν εθελοντές αυτοί. Και επομένως να σας πω τι έργο επιτελέσαμε με αυτή την έρευνα, κυρίως με τις μανάδες που συμμετέσχουν, 14 με 16. Και λίγο πριν τις ε, προεδρικές εκλογές έγιναν αυτά και οπότε ε, κατά κάποιο τρόπο ε, λάβαμε υπόψη τη ρόλο της οικογένειας, είχαμε αυτές τις αλλαγές τότε, και γι' αυτό και τελικά αποσύρθηκα από αυτή την αποστολή. Παρ' όλα αυτά ε, είχαμε έναν ευρωπαϊκό φορέα που μου ζήτησε να κάνω κάποια έκθεση ε, για το ότι πετύχαμε ποιοτικά και ποσοτικά και είχαμε 450 τέτοιους νέους για δύο γενιές διάφορες ε, μεταβλητές, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, ιστορικό της οικογένειας και γι' αυτό θα σας μιλήσω. Επίσης έκανα άλλες δύο εκθέσεις που δημοσιοποιήθηκαν ε, στο website του πράκτησης όσον αφορά την ριζοσπαστικοποίηση αυτών των 450 νέων. Όλα αυτά με τη βοήθεια της οικογένειάς τους για το θέμα του πώς θα σταματήσει η ριζοσπαστικοποίησή τους και 80% τα καταφέρανε και στη συνέχεια έχουμε κάποια στατιστικά ούτω ώστε να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί του κινδύνου, της προστασίας ε, και όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν συντόμως. Να επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας στο εξής θέμα. Στις οικογένειες, τους γονείς, τις μητέρες έχουμε 66% των ε, γυναικών ε, από τις 450 οικογένειες, 12 με 25 ετών ηλικίας και 15 και 12 ε, αγόρια και κοριτσιά αντιστοίχως οπότε είναι σημαντικό στοιχείο αυτό ε, επίσης διευκρινίζω ότι σε αυτό το δείγμα έχουμε 43% ε, οικογένειες ε, με αραβική καταγωγή Οι υπόλοιποι έχουν προσιλητιστεί, 43% είναι αυτοί, 50% από την μέση τάξη. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε καλύπτονται περισσότερο οι ε, μεσοαστικές οικογένειες παρά οι οικογένειες εργατικής τάξης. Και είπαμε, είναι για του για κορίτσια, ε, γιατί δεν βλέπουμε κάποια μεταβλητή ούτως ώστε να πούμε ότι αυτοί πρόκειται να ριζοσπαστικοποιηθούν. Τελικά στη ριζοσπαστικοποίηση οδηγεί πλειάδα μεταβλητών. Δηλαδή δεν είναι μια στιγμιαία κατάσταση, είναι μια ολόκληρη διαδρομή η ριζοσπαστικοποίηση. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί που τους επιστρατεύουν ε, το κάνουν από το ίντερνετ και αυτό που κάνουν είναι πολύ διάστατο, ε, κυρίως για τους ε, ανηλίκους, ε, ποντάρουν στην συναισθηματική φόρτιση, χρησιμοποιούν τον φόβο, στην έλλειψη εμπιστοσύνης, στη μη κοινωνικοποίηση, γιατί αυτοί οι νέοι πια δεν πιστεύουν στην κοινωνία, στον νόμο και θεωρούν αυτοί που τους επιστρατεύουν ότι θα τους πείσουν ότι πρέπει να πιστεύουν στον ε, θεϊκό και στον ανθρώπινο νόμο. Και έτσι αποκόβονται από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η αφετηρία της διαδρομής που οδηγεί στη ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό κάνουν οι στρατολόγοι, ας πούμε. και τους αναδεικνύουν, τους πλαισιώνουν και τους αγαπάνε κατόπιν στην ριζοσπαστική ομάδα. Προσπαθούν να αυτοκαθοριστούν, οι άλλοι γίνονται εχθροί, υπάρχει δεσπιστία, ε, αλλάζει μετά, γίνεται κάπως παρανοϊκή η άποψη των υπόλοιπων κόσμο, θεωρούν ότι αφού είναι έτσι η κατάσταση, τότε βρίσκονται σε νόμιμη άμυνα και οδηγούνται στην χρήση της βίας. Για να δούμε τα εξή τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, οι μανάδες είναι στην κατάλληλη θέση. Οι μανάδες μπορούν να επισημάνουν όλα αυτά, τις ε, συνέπειες από αυτή τη διαδικασία στρατολόγησης, από όλη τη ρητορική των τζιχαντιστών. Οι νέοι φοβούνται ότι προέρχεται από τους άλλους ανθρώπους μετά από αυτά που έχουν ακούσει από τους τζιχαντιστές. Και τελικά ε, συσχετίζουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Να, μονοθεϊσμός βασική αρχή του Ισλάμ. Επομένως, να τη, η βάση της στρατολόγησης είναι και πάλι ο φόβος. Επίσης, ε, κατόπιν, υιοθετούν την ε, τακτική της ρήξης. στέκονται κατά τις οικογένειες, σκίζουν τις φωτογραφίες. Γίνεται κάτι σαν Θεός και ο φωτογράφος. Καταστρέφουν τα αγάλματα. Δεν θέλουν να πάνε πια στο σούπερ μάρκετ, στο ΟΣΑΝ και μερικοί δεν παίρνουν καν το μετρό γιατί θεωρούν ότι ακόμα και ένας πλανόδιος μουσικός που παίζει μουσική και αυτός ότι είναι κάτι σαν Θεός. Να, επομένως τα καμπανάκια κινδύνου, τι μπορεί να δουν οι γόνιες στην καθημερινή ζωή επίσης όσον αφορά την απορριτσοσπαστικόποίηση. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία πάλι οι πιο κατάλληλη για να φρενάρουν αυτή τη διαδικασία είναι οι μανάδες. Πάντα για αυτή την προσέγγιση, την συναισθηματική φόρτιση του άγχους, του στρες, του, του, φόβου. Θα επανέλθουμε σε αυτό όμως ε, αργότερα για να καταλάβουμε το σύνολο της διαδρομής. Α, βλέπετε τώρα αυτή τη διαφάνεια, αλλά, είναι άχρηστη γιατί τα γράμματα είναι πολύ μικρά και δεν βλέπετε τίποτα. Σε αυτό το σλάι τέλος πάντων εγώ εξηγώ ότι με αυτή την προσέγγιση δημιουργούν κάτι σαν παράνοια τους νέους. Αυτοί θεωρούν ότι βρίσκονται σε νομιμή άμυνα και οι στρατολόγοι τελικά ε, ατομικοποιούν αυτή την ε, ε επιστράτευση, ε, τη στρατιωτικοποίηση, και υπάρχει διαφορά μεταξύ Τζιχάτ και Αλκάιντα γιατί τώρα το Ισλαμικό κράτος προσαρμόζει την ιδεολογία σε κάποιου είδους ε, συναισθηματικές και γνωστικές φιλοδοξίες ούτως υπήν του κάθε νέου. Υπάρχει επομένω εξατομικευμένη μεταχείριση και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερο υποκύπτουν σε αυτή την ε, υπόσχεση της αναγέννησης του κόσμου, ενώ τα αγόρια λένε ε, περιορίζονται στην ατομική αναγέννηση, αν μπορούμε έτσι να τα πούμε χονδρικά. Όμως υπάρχει πάντα αυτή η εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Υπάρχει διαβροποιημένη χρήση κινήτρων σύμφωνα με τα ιδανικά του καθενός. Και Υπάρχει αυτή η υπόσχεση προστασίας προς ε, κάποιους που έχουν υποστεί σεξουαλική βία, αλλά αυτό έχει κουκουλωθεί. Και έτσι προκύπτει και κάποιο είδους υπόσχεση εκδίκησης ε, για όποιον έχει υποστεί τέτοια πράγματα και οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση. Σύμφωνα με τις ερευνές μας, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να καταλαβεί κανείς τι υποσχέσεις έχει δώσει ο τζιχαντιστής για πώς τον ε, ήλκησε, πώς, το, τσίμπησε στο, στο, του τζιχαντιστή ο νέος. Άρα πρέπει να δούμε τι υποσχέσεις δόθηκαν. Ε, ε, πάλι οι γονείς και κυρίως η μάνα μπορεί αυτό να το διακρίνει και να μας τα καταγγείλει. και πώς έκανε τα πρώτα βήματα ο νέος προς αυτήν την ιδεολογία. Έχουμε τέσσερις προσεγγίσεις. Είπαμε πρώτα-πρώτα την συστηματική φόρτιση, τον φόβο, ε, το ότι τώρα ότι εντάσσεται σε ένα καινούργιο κύκλο, καινούργιες κοινωνικές σχέσεις, ε, το, το μαύρο άσπρο, άλλη οπτική για τον κόσμο και αυτό ανεξάρτητα από το τι παρελθόν είχε ο κάθε νέος, αν είναι μουσουλμάνος, χριστιανός ή άθεος. Τώρα, για να δούμε πάλι την επόμενη διαφάνεια που πάλι δεν την ε, διαβάζετε μικρά τα γράμματα, είναι το ότι τελικά οι γονείς έχουν ε, την αντίθετη προσέγγιση. Είπαμε τι κάνουν οι τζιγκαντιστέ. Η μάνα από την άλλη μεριά αυτό το οποίο κάνει είναι να έχει αυτή μια συναισθηματικά φορτισμένη προσέγγιση ε, η οποία οδηγεί στο πώς θα ξαναδώσει την ε, εμπιστοσύνη που χάθηκε. Η μάνα. Η μάνα είναι στην πιο κατάλληλη θέση ούτως ώστε να πλαισιώσει το παιδί και να το ξανααναδείξει η είπε. À Υποσχέσεις. Επομένως, από την ε, τζιχαντιστική ρητορική υπο, υποσχέσεις σε σχέση με την ε, κοινωνία, με το κοινωνικό συμβόλαιο. Οπότε, για να δούμε τώρα Τι μπορεί να κάνει η μάνα. Η μάνα έχει επεξεργαστεί αυτό το οποίο το ονομάζουμε ε, το, το πρότυπο του Προύστου. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν την ε, θεωρία, οι μανάδες που έχουν ενεργήσει με επιτυχία εφαρμόζουν αυτή την μέθοδο και είναι το 60% αυτό της δουλειάς που πρέπει να γίνει για να αποσυνδεθεί, να αποστασιοποιηθεί ο νέος από την κατάσταση. Και ο τζιχαντιστής, ο στρατολόγος έχει κόψει τους παλιούς συναισθηματικούς ε, δεσμούς και επίσης έχει εντάξει τον ε, νέο σε υποκατάστατη κοινωνική ομάδα και του έχει δώσει την ψευδέστηση ότι ανήκει σε κάποια μυθική ομάδα ότι, που είναι ανώτερη, που είναι ε, άγια σχεδόν και ε, του έχει δημιουργήσει ενοχές ο τζιχαντισμός για την ευχαρίστηση οπότε οι μανάδες προσπαθούν να ξαναγυρίσει στο παρελθόν το παιδί, να ξαναγυρίσει το σώμα του ούτως υπήν και να ξανεκτιμήσει τις μικρές χαρές της ζωής. Να ξαναθυμηθεί τα μικρά πράγματα, τα μικρά ορόσημα της παιδικής του ηλικία. Όλα τα οποία προηγήθηκαν πριν υποστεί αυτήν την αναισθησία πριν ε, απομακρυνθεί από τους... Ε, δηλαδή το αγαπημένο του γλυκό, την αγαπημένη του μουσική, ε, ό,τι ό,τι μικροπράγματα αγαπούσε. μια Εβραία του έδειξε του παιδιού ένα βίντεο από την παιδική του ηλικία και έτσι προκλήθηκε η συναισθηματική αντίδραση στον νέο του θύμισε το παρελθόν του. Κάτι το οποίο είχε σχέση με το σώμα του, με την προσωπικότητά του, ούτω ώστε να σπάσει αυτού του είδους το, το, το, κουκούλι που έχουν φτιάξει οι τζιχαντιστές ε, αυτού του είδους η, ε, η άρνηση της ανθρώπινης ιδιότητας γιατί για τους τζιγαντιστές δεν υπάρχει το άτομο, υπάρχει η ομάδα. Να λοιπόν πώς γίνεται αυτή η αποσύνδεση, πώς γίνεται αυτή η άπορη ζωσπαστικοποίηση. Οπότε ξαναβρίσκεται τον εαυτό του ο νέος. Είχαν ξεχάσει το σώμα τους, είχαν ξεχάσει τη μουσική τους και όταν ξανακούσαν βάλαν τα κλάματα κάποια αυτά τα παιδιά. Βλέπουμε επομένως κάποιες στατιστικές και λέμε ότι εκεί που δεν πήγαμε καλά ήταν 20% των ριζοβαστικοποιημένων. Και επίσης εκεί είχαμε 35% ανηλίκους και 65% ενήλικες από αυτό το 20% αποτυχίες. Να, αυτή είναι η μέθοδος η προύστια. Αυτό η οποία βέβαια κυρίως αφορά είπαμε τους ε, ανηλίκους γιατί οι ενήλικες πια μένουν μόνοι τους απομακρυσμένοι από τους γονείς τους και τελειώνω με κάποιες συστάσεις. Πιο εύκολη είναι η δουλειά μας με τα κορίτσια παρά με τα αγόρια. Αλλά δεν είναι θέμα φίλου, ξέρετε. Συμφωνώ με τις αναλύσεις μας, τα κορίτσια ευτυχώς ε, έχουν υπέρ τους αυτό το ακριβώς το ότι είναι οι γυναίκες. Δηλαδή αυτού του είδους η δογματική πυθός έχει πιάσει τόπο στα αγόρια περισσότερο παρά στα κορίτσια δηλαδή με ακριβώς τις ίδιες πράξεις, αντιμετωπίζεται διαφορετικά το αγόρι. Και δίνεται βάρος στην αστυνομική αντιμετώπιση του ριζοφαστικοποιημένου αγοριού παρά του κοριτσιού. Και λέμε ότι μετά τον πόλεμο η αντιφασίστες περιγράφουν τον ναζισμό ως μια επίθεση προς το άτομο και την οικογένεια. Και η αποκατάσταση ε, έγινε με την δημιουργία εκ νέου των οικογενειακών δεσμών. Αυτά γίνανε με αυτούς τους ε, Γάλλους ε, που είχαν προσιλητιστεί και πήγανε σε Ιράκ και Συρία δεν θα πρέπει αυτομάτως κανείς να υποψιάζεται τις οικογένειες. Δεν είναι κάτι το συστηματικό, κάτι το αυτονόητο το ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα παιδείας με τους ε, ριζοσπαστικοποιημένους. Οπότε το να δίνουμε την ε, σκητάλη της ευθύνη στους γονείς και κυρίως ε, στις ε, μανάδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να παρακάμψουμε ε, το, την κοινωνική πτυχή του θέματος. Και οι οικογενειακές ρήξεις δεν διευκολύνουν την έξοδο των ανηλίκων από την ζωσπαστικοποίηση Και όταν υπάρχει εξτομικευμένη διαδικασία σβαστικοποίησης, τότε θα πρέπει επίσης να είναι εξοδομικευμένη και η προσπάθεια της αποσύνδεσης του νέου από το τζιχαντισμό. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή της γυναίκας και δεν θα πρέπει να έχουμε συστηματική δημιουργία ρήξης Έχουμε ειδική ψυχομετρία, έχουμε επίσης ε, ειδικού επιστήμονες που χρησιμοποιούν όλες αυτές τις μεθόδους και έτσι να μπορεί να είναι μια σύμμαχος η μητέρα. Αυτό είναι το 60% της ε, δουλειάς της απόρριζος παστικοποίησης. Και σας ευχαριστώ. Thank, ε, you very much, Ms. Bozar, for your Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντούνια Μπουζάρ για αυτήν την παρουσίαση και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Τζιλ, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Παρακαλώ. Ε, bueno, me gustaría, ante todo... Καλημέρα σας. Πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε και να ξεκινήσω με μία μικρή διευκρίνηση διότι μιλούμε για τις γυναίκες ως μια κοινωνική ομάδα γιατί μιλούμε για ένα κομμάτι της κοινωνίας, μιλούμε για την πρόληψη, μιλούμε για κάποια μέτρα τα οποία προτείνονται σε επίπεδο πολιτικής, παιδείας για τις ακτιβίστριες. και λέμε ότι έτσι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση της γυναίκας. Ε, entonces, me Η αυτή γυναίκα λοιπόν είναι ακτιβίστρια, μπορεί να είναι ψυχολόγος και πήραμε πάρα πολλές ε, συνεντεύξεις για να δούμε ποιο είναι το προφίλ αυτών που είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί Μπορούν και οι συνάδελφοι τώρα να σας τα εξηγήσουν περισσότερο και θα, αυτές οι γυναίκες εξετάσαμε τη δουλειά κάνουν, σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν και για αυτό το βιβλίο. Να σας πρώτα πρώτα τι έγινε, τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. La palabra a las madres para que ellas mismas denunciasen la visión de, de la problemática que ellas vivían. Για να δούμε επομένω ποια είναι η προβληματική όσον αφορά την καθημερινή τους ζωή. Τι πρόβλημα υπάρχει όσον αφορά την πρόληψη. Τι γίνεται με αυτές τις καταγγελίες από το 12 μέχρι το 13. Τότε δεν υπήρχε κανένας είδους εκστρατεία, τίποτα για τα ε. Σήμερα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, να παρακολουθήσουμε την ταχύτητα της εξέλιξης με κάποιο είδους ε, ενιαία μέθοδο. Πάμε για τις ε, μανάδες, είπαμε τα πανεπιστήμια πώς προσπαθήσανε να βρουν κάποιον κοινό παρονομαστή. Προσπαθήσαν να αποσυνδέσουν ε, αυτά τα άτομα από την πραγματικότητα και να μπουν στον κόσμο της βίας. Οπότε είναι πάρα πολύ ε, λάθος να πέσουμε σε εντετερμινισμό όσον αφορά το ότι για όλα είναι θέμα ε, μια κοινωνική αντιμετώπιση, ένα ρατσισμός ε, όσον αφορά τη, την τακτική δηλαδή των τζιχαντιστών. Μιλούμε επομένω για αυτές τις μανάδες. Μιλούμε για το ότι σήμερα είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν. από αυτές τις ε, οικογένειες ε, από την Ισπανία και επίσης κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου οι περισσότερες από αυτές τις μανάδες και υπήρχαν και αδελφές και αδελφοί στην υπόθεση. Και όταν φύγανε να πάνε Συρία ή Ιράκ, αυτοί οι νέοι στις περιπτώσεις που είδα, η, η ριζοσπαστικοποίηση εντάθηκε εκεί στην εμπόλεμη ζώνη. Συνεχίστηκε κάποιο είδους σχέση, σύνδεσμος σχεδόν πάντα με αδελφή, αδελφό μάνα και όχι τόσο με τον πατέρα. Θεωρήθηκαν σαν ένα αντικείμενο στο οποίο εφάρμοσαν οι τζιχαντιστές τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης. Και το κάνουν και σε γυναίκες όπως και σε άντρες. Έχουμε και εκείνη την αποτυχημένη τρομοκρατική απόπειρα από δύο Γαλλίδες ε, στη Νότρο στο Παρίσι και υπάρχει το στερεότυπο ότι η γυναίκα είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον άντρα και αυτό στερεότυπο είναι Οπότε οι τζιχαντιστές όμως απευθύνονται και σε νέους και σε νέες για να τους στρατολογήσουν. Και θεωρούν ότι η μουσουλμάνα που φοράει το, ε, το, το τσαντόρ ας πούμε και είναι υποτακτική στον άντρα της μπορεί να ισχύσει το ίδιο σε σχέση με το Ισλαμικό κράτος. Λέμε τώρα για τους Ευρωπαίους που στατρογούνται στην Ευρώπη. home grown. Είναι διαφορετική η κίνδυνη ανάλογα με το φύλλο. Έτσι όμως υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμήσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός συναντήσεις, συνεδρίες, Ε, δημιουργία ζευγαριών, προπαγάνδα στο ίντερνετ και αυτός ο μηχανισμός γίνεται από και για τις γυναίκες πολλές φορές. οι συναδέλφοι σας μπορεί να σας τα εξηγήσουν. Έχουν μελετηθεί διάφορες συζητήσεις μέσω των ε, κοινωνικών δικτύων. Και βλέπουμε ότι υπάρχει βία ή απειλή βίας που είναι ανατριχιαστική έναντι των γυναικών. Γι' αυτό σας έλεγα για αυτή την τρομακτική ενέργεια που τελικά χρησιμοποίησαν βουτάνιο, τελικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια, μια κοπέλα που είχε τρία παιδιά, 29 ετών και που κουβάλαγε το βουτάνιο. Και η ερευνά κατατείνει στο ότι αυτή η γυναίκα επιστρατεύτηκε από το ίντερνετ. Ήξερε βέβαια τις τεχνικές, ε, αλλά την στρατολόγησαν τέλος πάντων γιατί θεωρήθηκε ότι είναι λιγότερο επικίνδυνη από έναν άντρα για τη δουλειά. Και φυσικά όταν ασπαστούν την ιδεολογία του τζιχαντισμού είναι πιο εύκολο να πάρουν τα όπλα αυτά τα πρόσωπα. Άλλες περιπτώσεις. Ο Μαξίμ ε, επιστρατεύθηκε, στρατολογήθηκε τέλο πάντων στην Γαλλία. Παντρεύτηκε με μία μουσουλμάνα. Αυτή ήταν τζιχαντίστρια. Τώρα δεν θέλει να γυρίσει. Λέει η μάνα του γιατί ο πατέρας του δεν είναι εκεί και ήδη έχει κάνει ένα παιδί στη Συρία ο Μπερτράν το αντίθετο έχει πέντε παιδιά ήταν 19 ή 20 όταν ε, είχε ενδιαφέρον για τα πνευματικά ε, είχε ασχοληθεί και με τον βουδισμό πριν γίνει μουσουλμάνος. Οπότε και, όπως πολλά άλλα ζευγάρια πήγαν και οι δύο στην Συρία. Είναι αυτό το στερεότυπο που λέγαμε πριν. Είναι μια Βελγίδα. Δεν αν την έχετε ακούσει. Ο Ταρέκ είναι ο σύζυγός της, μένανε στο Σκαρμπέκ εδώ ήταν 18 και πήγε στη Συρία και μετά από δύο εβδομάδες σκότωσε τον σύζυγό της. Μπορούσε να γυρίσει αλλά δεν το έκανε. Κάθισε εκεί έξι χρόνια. Δεν θέλει να γυρίσει είναι μία από τις χείρες του Ισλαμικού κράτους. Όπως λέει η μητέρα της, δεν ε, μετανιώνει. Συνεχίζει να έχει επαφή η μάνα με την κόρη. Ξαναπαντρεύτηκε. Όπως πολλές από τις χείρες της ΝΤΑΕΣ. Α, να, να στα πω γρήγορα για να μην ξεχάσω τίποτα. Βλέπουμε ποια είναι η εμπλοκή των ε, γυναικών και αντίθετα από ό,τι σκέφτεται κανείς οι Ευρωπαίοι τζιχαντιστές ε, και οι γυναίκες τζιχαντίστριες δεν είναι ε, νοικοκυρές. Αυτές θέλουν να τις βάλουν, θέλει η τζιχάτ να τις βάλει κάπου μες στον κοινωνικό ιστό. Και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι λένε οι μητέρες, τι λένε για τη θέση τους στην κοινωνία, στα επαγγέλματά τους, για να δούμε πώς θα γίνουν οι διάφορες εκστρατείες πρόληψης. Μια νοσοκόμα, μια που δουλεύει στο Παρίσι για ανθρώπινους πόρους, για μια άλλη σε μεγάλα καταστήματα, μια καθαρίστρια λοιπόν και άλλη που δουλεύει στο Δημαρχείο του Παρισιού. Αυτά για το προφίλ των νέων, αλλά θα πρέπει να δούμε και το προφίλ των μανάδων, αν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην διαδικασία της πρόληψης. Τι θέσεις έχουν, ποιες είναι αυτές, ε, εμπλέκονται στη δημόσια ζωή, στον κοινωνικό ιστό, τι θέση έχουν. Καταδικάζουν αυτό που κάνουν τα παιδιά τους καταδικάζουν ότι έκαναν τα παιδιά τους στην ε, Συρία ή στη Γαλλία. Πολλές φορές όμως δεν έχουν τον εγκαίο χώρο, διότι θεωρήθηκε ότι είναι συνένοχες, συναυτουργοί ή ριζοσπαστικοποιημένες. Είτε ήταν μουσουλμάνες είτε όχι και δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Δεν έχουν μόνο στο περιθώριο. Είναι στιγματισμένες και φοβούνται. Και φοβούνται μην χάσουν και τη δουλειά τους. Όταν γίνει ό,τι έχει γίνει με το γιο τους, τον άντρα τους. Επίσης, είναι σημαντικό να προβληματιστούμε πώς θα μπορούν να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη αυτές οι μανάδες προς τις αρχές. Να σταματήσουν να φοβούνται την συνεργασία. Να έχουμε επίσης και κάποιες δομές όσο γίνεται πιο κοινέ στην Ευρώπη. Να δούμε ποιες είναι οι καλές, ποιες οι κακές ε, πρακτικές και να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτή την πρόληψη της ζωσοφαστικοποίησης. Τι γίνεται όταν δεν συνεργάζεται μία μάνα. Πολλές είναι αυτές που δεν συνεργάζονται. Είπα για τις αδελφές, τις νέες αυτές που εμπλέκονται, τα είπα στο βιβλίο και πέραν των ε, γνωστών οικογενειών τελικά είπαμε ότι δεν ξέρουμε και πάρα πολλέ οικογένειε που έχουν εμπλακεί έτσι. Πόσοι επομένω είναι οι οικογένειε που εμπλέκονται, δεν έχουμε, χάνουμε πληροφορίε, δεν ξέρουμε πού είναι αυτοί οι νέοι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με την ε, επιστράτευσή του. Είναι επομένω ε, κακά τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε ακριβώ γιατί από φόβο πολλέ οικογένειε δεν είπαν τίποτα φοβήθηκαν πως χάζουν τη δουλειά τους η σιωπή επομένω αυτών των ε, μανάδων εχθρότητα προς ε, τις κρατικές δομές. Στις γαλλικές φυλακές πρόκειψε... ότι ένας από, το, ένας από τους φόβους των ε, θεσμοφυλάκων είναι ότι υπάρχουν κάποια δίκτυα εκεί πέρα. Όταν πάνε οι μανάδες να μιλήσουν στα παιδιά τους, Υπάρχει αυτό το δίκτυο λοιπόν των οικογενειών και έτσι αυξάνεται αυτή η εχθρότητα προς το κράτος. Ε, το κοινό αυτών των οικογενειών είναι ότι είναι φυλακισμένο το παιδί τους. Ε, αυτό είναι το κοινό σημείο των μανάδων που ανήκουν σε αυτά τα δίκτυα. Η φυλακή είναι μακριά από το σπίτι τους. Και ε, επομένως υπάρχει κάποια κοινή προσπάθεια Πήγα στη Βόρεια Γαλλία πρόσφατα σε μια φυλακή και οι δεσμοφύλακε μου λέγανε 40, 40 ήταν αυτοί με του. μίλησα και είπανε ότι οι μανάδε του ήταν κοντά στα παιδιά του που είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί και είπαν οι δεσμοφύλακε ότι έρχονται κάθε εβδομάδα αυτέ οι μανάδε και εμεί θεωρήσαμε ότι και αυτέ είναι ριζοσπαστικοποιημένε. Όμω αυτό είναι στρεβλή οπτική, είναι ένα στερεότυπο. Οπότε χειροτερεύει τα πράγματα, ούτε βοηθάει την ε, πρόληψη. Χρειάζεται διάλογος. Ε, Είπαμε θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια και μετά την επιστροφή των νέων και δεν φτάνει η απορροζοσπαστικοποίηση. Ωραία λέξη είναι, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε να εγκαταλείψουν την εικόνα της βίας μέσα στην ε, οικογένεια. Να δούμε ποιος είναι στη φυλακή, τι κάνει ο μικρός αδερφός, αυτόν που είναι στη φυλακή. Η δυσπιστία προς τη φυλακή, προς το κράτος. Τι κάνει, δηλαδή τι είναι η φυλακή, ε, είναι μέσο για την ε, λύτρωση, τι είναι, απλώς ε, η παράταση της ε, άσχημης κατάστασης. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσετε σιγά σιγά. Σαράντα είναι αυτοί που εξέτσαν την ποινή του και θα αποφυλακιστούν τώρα. Οπότε διάλογος για την απολυσία του είναι κάτι το αναγκαίο, κάτι το επιτακτικό. Θα πρέπει η γυναίκα να εμπλακεί ε, σαν μάνα και όχι μόνο σε αυτό. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αλεξάνδρα Ατζήλ και θα ήθελα τώρα να δώσω τον το λόγο στην Κάρολα Γκαρσέα Κάλβου στην Ιωράλαλη στο πρόγραμμα για τον Παγκόσμιο για την παγκόσμια τρομοκρατία στο Ελκάνο Royal Institute. Ε, επειδή θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει στις 11, δεν θα σας δώσω πολύ χρόνο για να Μετά αφού θα ε, χρειαστεί συνέχεια να δώσουμε και συνέχεια το λόγο στους ε, συναδέλφους προκειμένου να σας θέσουν κάποια ερωτήματα, στα οποία συνέχεια βέβαια θα πρέπει να απαντήσετε. Οπότε έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας πω τι γίνεται με αυτές τις μελέτες που έχουμε στο Βασιλικό Ίδρυμα Ελκάνου. Όπως είπαμε για σήμερα το πρωί, όντως ο ρόλος της γυναίκας στις τρομοκρατικές οργανώσεις πολλές φορές υποτιμήθηκε και υπάρχουν κάποιες μελέτες που εμπειρικά προσπαθούν να προσεγγίσουν τον ρόλο των γυναικών ή τους ρόλους μέσα στην οργάνωση. Και βλέπουμε γιατί, από που προέρχονται αυτές οι γυναίκες και γιατί ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Έχουμε αυτές τις μελέτες. Επεξεργαστήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία στο Ελκάνο και έχουμε αυτές τις γυναίκες που έχουν καταδικαστεί στην Ισπανία. Το θεματολόγιο μας είναι κάπως φιλόδοξο σε σχέση με τον χρόνο που έχουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σύντομη, σύντομη. Και μετά να δούμε τι ερωταπαντήσεις. Να δούμε. Περί ομιλούμε. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν καταδικαστεί 117 πρόσωπα για δραστηριότητες σχετικές με την τζιγαντική τρομοκρατία. Από το 2012 έγινε τελευταία κινητοποίηση σε σχέση με τον πόλεμο στη Συρία και όλα αυτά από το Ισλαμικό κράτος. Από το 2004 που είχαμε τρομοκρατικές απόπειρες στη Μαδρίτη έχουμε ε, πόλεμο με αυτούς και είπαμε ότι έχουμε επίσης από τότε μια ομάδα τρομοκρατική που υπάρχει στην Αλκάιντα. Από το 2014 όμως καμία γυναίκα δεν συνελήφθη. Και στην ε, Μελίγια τότε συνελήφθη που προσπάθησε να περάσει στο Μαρόκο μια κοπέλα 14 ετών. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε 13 γυναίκες από όλους τους συλληφθέντες ή καταδικαστέντες. Όλα αυτά από εμπειρική μελέτη, επί τη βάση μιας βάσης δεδομένων. Όλα στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να τα βρείτε. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες που ασχολούνται με την τζιχαντιστική τρομοκρατία στην Ισπανία για να δούμε επίσης τι γίνεται μέσω αυτού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες που ασχολούνται και εμπλέκονται είναι νέες. Πιο νέες από τους αντίστοιχους άντρες. Βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια ότι αυτοί οι καταδικαστέντες έχουν μέσω χώρο ηλικίας 30 έτσι. Οι γυναίκες τέσσερα χρόνια πιο νέες. Στα 26 δηλαδή. Άλλη μεταβλητή, σημαντική για να καταλάβουμε τι είναι αυτές οι γυναίκες, είναι η οικογενειακή τους κατάσταση. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τους άντρες. Έχουν συνήθως οικογένεια οι άντρες. Οι γυναίκες, είπαμε, είναι νεότερες, αλλά συνήθως είναι ανήπαντρες, χωρίς υποχρεώσεις. Αυτή είναι η στρατηγική του Ισλαμικού κράτους. Τέτοιες γυναίκες ε, ελκύει, γιατί θέλει να τις πάρει και θέλει πέραν των όπλων να χρησιμοποιήσει τις γυναίκες για να κάνει κάτι σαν απικία για να μπορέσει το χαλιφάτο να επεκταθεί με την εγκατάσταση εκεί τέτοιων γυναικών. Άλλο εργαλείο που έχουν δηλαδή είναι το πώς θα εκπαιδεύσουν την επόμενη γενιά τζιχαντιστών τώρα. Για να δούμε πώς γίνεται αυτού του είδους η ένταξη στο τζιχαντιστικό κίνημα για αυτές τις γυναίκες. Εδώ λέμε ότι έχουμε την τρομοκρατία homegrown που αναπτύσσεται δηλαδή στις χώρες μας. Επειδή έχουμε πάρα πολλούς από δεύτερη γενιά εδώ, στο δείγμα, πάντως λέμε για κάποιες γυναίκες που γεννήθηκαν στην Ισπανία. Στη συνέχεια βλέπουμε για την ζωσπαστικοποίηση, για να καταλάβουμε το πώς γίνεται αυτή η διαδρομή, αυτή η διαδικασία. Από το 12 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Συρία, που μετά επεκτάθηκε στο Ιράκ, έχουμε την περίοδο 12 με 15 σε αυτά τα χρόνια είχαμε αυτή την κορύφωση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης το 14 ο Αλμπαγκντάντι προσπάθησε να μεταναστεύσει το Χαλιφάτο στο Χαλιφάτο δηλαδή να πάνε οι αυτές οι γυναίκες αφού μαζεύουν τα προγραμματά τους εκεί πέρα και είπαμε ότι ε, ήταν πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, τους έδωσε ένα όραμα ζωής, τους έδωσε μια ευκαιρία να αναπτυχθούν εκεί ως μάνες, ως γυναίκες και ως εγγυητές αυτού του οράματος αυτού που, που, που είχε ο Μπαγκδάντι. Και είπαμε ότι πολλές φορές αυτά είναι πιο αποτελεσματικά από τα όπλα τους, γιατί τους είπε πώς θα μπουν σε αυτό το οικοδόμημα που έφτιαχνε ε, και ότι έχουν ρόλο κλειδί σε όλα αυτά. Είπαμε ότι ξεκινάνε αυτή τη διαδικασία πιο νωρίς από τους άντρες 20 ετών περίπου, ξεκίνησαν όλα αυτά, πιο μεγάλοι οι άντρες. Δηλαδή ήταν γύρω στα 26 όταν έκαναν τα αντίστοιχα οι άντρες. Τώρα κάτι άλλο ενδιαφέρον. Η σημασία του ίντερνετ για την ριζοπραστικοποίηση των γυναικών. Οι περισσότεροι καταδικαστέντες ριζοσπαστικοποιήθηκαν σε μεικτό περιβάλλον. Ιντερνετικά και εκτός ίντερνετ. Σε άμεση προσωπική επαφή με τους λουδοσυπήν στρατολόγους. Οι γυναίκες περισσότερο μέσω του ίντερνετ. Να, το πόσο ωφελήθηκε το τζιγατιστικό κίνημα από το ίντερνετ για τις γυναίκες. Παλιότερα που οι γυναίκες λοιπόν δεν ήταν στο ίντερνετ, ήταν στην οικογένεια, γινόταν, προσπαθούσαν να μπουν μέσω της οικογένειας για να τις τατολογήσουν. Ήταν θέμα λοιπόν το πόσο μπορούσαν οι τζιγατιστικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση στο σπίτι, στο νοικοκυριό, στην οικογένεια για να στατολογήσουν αυτές τις γυναίκες. Αυτά γίνανε στην Ισπανία. Σημαντικά όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία αυτής της προσέγγισης ε, της ιντερνετικής, τα κοινωνικά δίκτυα, κάθε είδους, οι ε, γυναίκες μαζί με άλλους, πάντοτε που θα δούμε στη συνέχεια, επίσης τα messengers, τα διάφορα, τα κινητά και το ίντερνετ είπαμε, τα blogs, όπως είπε κάποια στιγμή και η συνάδελφος η Αλεξάνδρα. Τώρα όσον αφορά το περιβάλλον εκτός ίντερνετ. Και αυτές τις μεθόδους να μην τις υποτιμούμε γιατί εκεί σε ιδιωτικές συναντήσεις είχαμε στρατολόγηση σε πολιτιστικά κέντρα ή γύρω από αυτά στο περιθώριο επομένω των πολιτιστικών Ισλαμικών κέντρων εκεί πολλά συζητιούνται και οι πολιτικοί μαζί με τα άλλα συνεχίζουμε τώρα και να δούμε Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως είπαμε πριν, στη βάση δεδομένων μας, δεν έχουμε καμία γυναίκα που ριζοσπαστικοποιήθηκε μόνη της, μέσα στο σπίτι, μόνη της. Είχε την προπαγάνδα, την σαλαφιστική και έτσι προσχώρησε σε τέτοιες βίες δραστηριότητες. Πάντα γινόταν όχι μόνη της, αλλά με άλλες, με άλλες κοπέλες. Και έτσι κατέληξε στην ιδεολογία της βίας, στην ιδεολογία του μαύρου και του άσπρου, στο ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Πολύ σημαντικό αυτό για την ριζοσπαστικοποίηση. μαζί με άλλες. Επομένως, που πήγαν τελικά στο Χαλιφάτο ή έμειναν στην χώρα τους, έμειναν στην Ισπανία και ψάχνανε άλλες γυναίκες για να τις ατολογήσουν και να τις στείλουν στο εκεί, στο μέτωπο. Και ακτιβιστές και άνδρες που ήταν στην ε, οργάνωση. Αυτοί οι άντρες ε, τραβούσαν τις γυναίκες γιατί ε, ήταν πολλοί άντρες όπως λέμε, είχαν την εμπειρία, τέτοια εικόνα. Στο Ελκάνο επίσης επισημάναμε ότι υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ αυτών των ε, ανθρώπων που καταδικάστηκαν με άλλους. Με άλλους, με αυτούς που λέμε foreign fighters, τους ξένους μαχητές. Πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται οι τρομοκρατικές ομάδες. Να, στο Ριπόλ. Υπήρχε, υπήρχαν και ξένοι μαχητές που φέρνανε άλλο κόσμο. Πιο μικρούς, γυναίκες κλπ. Να μην ξεχνούμε όμως ότι πάντοτε η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτά μια που δεν έχω άλλο χρόνο και να απαντήσω σε ό,τι ρωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Σαλότη Ζαξόν ε, που είναι υψημόμαθμη εμπειρογνώμονα σε ζητήματα φίλου στο EAS. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε τους διοργανωτές αυτής της ε, πολύ σημαντικής ε, συνάντηση ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις προηγούμενες ομιλήτριες για τις πολύ σημαντικές παρεμβάσει που έκαναν σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διάσταση της πολιτικής και το τι κάνουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Επιτρέψτε μου καταρχήν ε, να σας πω ότι δεν μπορούμε να αποτρέχουμε σε ό,τι αφορά ε, κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να λύσουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα ενισχύαμε τα στερεότυπα που ήδη φύστανται και στα οποία αναφέρθηκαν οι προηγούμενες ομιλήτριες. Επίσης θα πρέπει να ε, εξετάσουμε προσεκτικά τον τρόπο σκέψης μας προτού τοποθετηθούμε. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι αν θέλετε, να είμαστε ουδέτεροι και να μην προτρέχουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία ορισμένες φορές επιδεκνύονται υπερβολικά και τα οποία δεν είναι ουσιαστικά αληθή, γιατί έχουμε δει δηλαδή να υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Άρα λοιπόν εδώ στη σημερινή συζήτηση αναφερόμαστε στο ρόλο των γυναικών ε, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά να αναφέρουμε εδώ ε, και τους πολυάριθμους ρόλους τους οποίους παίζουν οι γυναίκες, όχι μόνο ένα ή δύο. Και επίσης να αναφέρουμε και την διάσταση ε, της γυναίκας σε διάφορα επίπεδα, γιατί για παράδειγμα το φύλλο δεν έχει να κάνει για παράδειγμα μόνο με τον άντρα ε, και την γυναίκα, αλλά έχει να κάνει και με την θηλυκότητα ή την ερενοπότητα, πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τον άντρα και τη γυναίκα ως σεξουαλικά όντα. Εντάξει από εκεί και μετά να πω αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ο κόσμος σας είναι επικίνδυνος και τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν ένα από τους εκείρους εταίρους μας σε ό,τι αφορά την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης ως προς τον τρόπο εργασίας μας. Ήδη ανέφεραν και ε, εκείνα ε, το 2017 ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε μια διπλωματία για την ειρήνη καθώς και οι συγκρούσεις μας ε, καθίστανται όλο και πιο περιπλοκές και λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με αποτέλεσμα βέβαια η ριζοσπαστικοποίηση και η θεωρητική μίσους και η βία γενικά να εξαπλώνονται. Ε, παρότι λοιπόν ε, γενικά ε, η Μπόκο Αράμ, η Αλσαμπάντ ε, το Ισλαμικό κράτος είναι τέτοιου είδου τρομοκρατικές οργανώσεις του Ισλάμ στις οποίες έχουν εστιάσει ιδιαίτερα τα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και περαιτέρω οργανώσεις οι οποίες έχουν ανακύψει σε ε, διάφορα άλλα μέρη. Για παράδειγμα, στον Καναδά και στι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν μελέτε που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποια μιλήσια, κάποιε δηλαδή παραστατικέ ομάδε, οι οποίε προωθούν, για παράδειγμα, την ανωτερότητα τη λευκή φυλή και οι οποίε εξαπλώνονται ολοένα και ταχύτερα ε, ταυτόχρονα στη Μιαμάρα, στη Στρι Λάνκα και στην ε, Ταϊλάνδη υπάρχουν Αντίστοιχε ριζοσπαστικέ οργανώσει, οργανώσεις, ενώ στην Ινδία οι ριζοσπαστικές ακραίες συντουιστικές οργανώσεις ε, ενισχύονται όλο και περισσότερο. Άρα λοιπόν όλε αυτέ οι οργανώσει, όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεν δηλαδή παρατηρούμε αμυγό θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση. Η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να είναι και πολιτική. Και συχνά είναι στενά συνδεδεμένη η θρησκευτική με την πολιτική. Και παρότι αυτές, αυτά τα ρεύματα αυτές τις οργανώσεις ε, δείχνουν να είναι διαφορετικές, ε, συχνά ακολουθούν τις ίδιες κατευθύνσεις, δηλαδή ε, προβολή μιας ταυτότητας και την άσκηση πιέσεων προκειμένου κανείς να επιλέξει συγκεκριμένη ταυτότητα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εθνότητα ή τη θρησκευτική. Επίσης επιβάλλουν συγκεκριμένες περιγραφές σε ό,τι αφορά την αρνοπότητα και τη θηλυκότητα που έχουν αντίκτυπο στο πώς γίνεται αντιληπτός και πώς αναμένεται να συμπεριφέρεται ο άντρας και η γυναίκα σε ό,τι αφορά του ρόλο και επίσης αυτές οι οργανώσεις συνηθίζουν να ε, ρίχνουν το, ε, το, το, την ευθύνη για προβλήματα στους άλλους και αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες. Ε. Και από εκεί και μετά το νόμισμα, αν θέλετε, στην πολιτική οικονομία αυτών των οργανώσεων συχνά είναι η γυναίκα και η θελικότητα που σας είπα δεν είναι πάνω με ό,τι έννοιες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό ο οποίος ε, σχετίζεται και με την αυξανόμενη μετανάστευση και την ε, ε, στο Ισλάμ ε, σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αυτό που εκλαμβάνουν οι μετανάστες από την ε, Συρία ε, σε σχέση με την υποδοχή τους από τις δυτικές χώρες είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται για παράδειγμα με την θυματοποίηση ε, και την απώλεια της ταυτότητας και την και τέτοιου είδους ε, ε, όλες αυτές, όλη αυτή η αίσθηση ε, δημιουργεί περισσότερη δικαιολόγηση σε ό,τι αφορά την άσκηση βίας έναντι των άλλων και έχει αναφερθεί για παράδειγμα και από τον Μερτή Χάτσον ο μεγάλος αριθμός νέων ανδρών που συμβάλλει στην ακραία ριζοσπαστικοποίηση και στις ευβίες σύγκρουσες. Όλες οι ακραίες οργανώσεις αποκλείουν όλους όσους δεν προσυπογράφουν τις ίδιες αξίες ενώ εξέρουν τους αυτούς τους και με αυτόν τον τρόπο βέβαια ε, αφαιρούν τον ανθρώπινο χαρακτήρα από εκείνους τους οποίους ε, ε, αποκλείουν δημιουργώντας ακριβώς έφορο έδαφος για περισσότερη βία ε, όλο ένα και περισσότερες ε, μελέτε και βιβλιογραφία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ένας ε, και μόνο λόγο για αυξανόμενη διακαιρισσοσπαστικοποίηση. Υπάρχουν δηλαδή και με την πάρδο του χρόνου διαφορετικές ε, παράμετροι οι οποίες δίνουν κίνητρα και σχετίζονται με τις, την πολιτική διακυβέρνηση, τι οικονομικέ και κοινωνικές συνθήκες και δημιουργούν ακριβώς τις βασικές αιτίες τη ρισοσπαστικοποίηση. Και εμεί από την πλευρά της εξωτερική Εξωτερικής ε, το θεωρούμε ως εξαιρετικά σημαντικό να εξετάζουμε ακριβώς αυτές τις βασικές αιτίες της ριζοσπαστικοποίησης ε, για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις. Και θα πρέπει να εργαστούμε σε όλα αυτά τα επίπεδα ταυτόχρονα για να κάνουμε τη διαφορά. Ε, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών γνωρίζετε πως έχει οθετηθεί εμφατικά αυτός ο στόχος δηλαδή της καταπολέμησης του εξτρεμισμού και τις ριζοσπαστικοποίησης ε, και υπάρχει και ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ε, ε, ουσιαστικά θέτει το μοντέλο σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των εθνικών σχεδίων δράσης και Εκείνο που αναφέρεται εκεί είναι ότι το empowerment, δηλαδή η απόδοση αυτοεξουσιότητας στις γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. γιατί παρότι οι γυναίκες ορισμένες φορές παίζουν κάποιο ρόλο στις βίες ακραίες οργανώσεις, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονό ότι στι κοινωνίε εκείνε όπου υπάρχει περισσότερη ισότητα μεταξύ ε, των δύο φύλων υπάρχουν λιγότερα φαινόμενα ε, ε, βία και ριζοσπαστικοποίηση. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να μα δείξει έναν μακροπρόθεσμο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο στο να επιτύχουμε περισσότερη αυξησιότητα για τι γυναίκε και περισσότερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια είναι πολύ σημαντική και η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση για παράδειγμα με την εξάλληψη της ένδυας ε, και την δημιουργία ε, δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών. Πρόκειται λοιπόν εδώ για εργαλεία ε, τα οποία παρακολουθούμε στενά στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, αποκινούμε άλλες οργανώσεις εταίρους σε πολυμερές επίπεδα, εκ των οποίων βέβαια είναι σημαντικότερο ο ΙΕΛ, από εκεί και μετά και άλλες. Και να αναφέρω εδώ, για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ, τον ΟΣΑ, την Αφρικανική Ένωση, συγγνώμη, την ΟΑΣΕ, την Αφρικανική Ένωση, τι διάφορε οργανώσει τη Λατινική Αμερική και ούτω καθεξή. Ε, αντιμετωπίζουμε κοινέ προκλήσει με αυτέ τι οργανώσει, ε, μπορούμε να άλληλο υποστηριχτούμε. Η ριζοσπαστικοποίηση αποτέλεσε πάντοτε βέβαια το σημείο στο οποίο ε, συγκρούονται διάφορε ιδεολογίε και ρεύματα σκέψη προκειμένου να επιβάλλουν το δικό του τρόπο σκέψη στην κοινωνία και βλέπουμε πω αυτέ οι, οργαν... οι οργανώσει ριζοσπαστικοποίηση χρησιμοποιούν τέτοιου είδου πλατφόρμε, είτε είναι θρησκευτικέ είτε είναι πολιτικέ. Γιατί βέβαια πάντοτε χρησιμοποιούν και υπό πολύ έξυπνο, τρόπο το φύλλο ως ε, εργαλείο. Σε αυτό προσπαθούν να κάνουν Δηλαδή το χρησιμοποιούν ακριβώ, χρησιμοποιούν τη διάσταση του φύλου ακριβώ για να συγκεντρώσουν περισσότερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά ε, τι ε, ακραίε ιδέε του, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ε, την ε, προσευχή, την δημιουργία περισσότερη σύγχυση, σε ό,τι αφορά την ε, θρησκεία, αλλά και ιδιαίτερα αυτό που παρατηρούμε τώρα τελευταία είναι η αίσθηση ταυτότητα, η δημιουργία θυμού σε ό,τι αφορά τι αδικίε και ό,τι καθεξή. Άρα λοιπόν, ε, με βάση την ε, συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το σεβασμό της αρχής ισότητας μεταξύ όλων, αυτά είναι όλα βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους προωθούμε ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση για τη βία. Αλλά αυτές οι οργανώσεις γνωρίζουν καλά πώς να χρησιμοποιούν τα δίκτυα κοινωνική δικτύωση προ όφελό του. Και γνωρίζουμε πω αυτά τα δίκτυα, παρότι φυσικά επιφέρουν πολλά πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολύ αρνητικούς και καταστροφικούς σκοπούς. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς από τη δική μας πλευρά. Ε, συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις όπως είπαμε. Ε, και ναι, έχω κατά ότι πρέπει να ολοκληρώσω πρόεδρε και ότι μου μένει 1,5 λεπτό. Ε, για παράδειγμα, μαζί με την Αφρικανική Ένωση πέρυσι υπήρξε μια κοινή δήλωση ως προς τον τρόπο καλύτερης αντιμετώπισης ε, ε, ε, του βίου και της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με πολυμερείς οργανώσεις και αυτή την περίοδο ε, ενημερώνουμε ε, τον ρόλο των γυναικών σε ό,τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να παίξουν και στι περιόδου μετά από τι σειράξει και υπάρχει μια εσωτερική εδώ εφαρμογή και εξωτερική εφαρμογή. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τα όσα κάνουμε εμεί στα δικά μα κράτη-μέλη, αλλά και με το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τρίτε χώρε. Κάτι ακόμα το οποίο συντάσσεται αυτή την περίοδο και για το οποίο θα θέλαμε να υπάρξουν συμπεράσματα του Συμβουλίου πριν από τα τέλη του 2018. και το οποίο θα αναφέρεται και με περισσότερη έμφαση μέσα στη νέα πολιτική είναι η ε, ε, καταπολέμηση και η πρόληψη ε, του βιοεξτρεμισμού και αποτελεί φυσικά και στοιχείο μέσα στη συγκεκριτική ατζέντα το θεματολόγιο για τις ε, γυναίκε ε, σε ό,τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια. Άρα λοιπόν εδώ διαπιστώνουμε ότι κατανοούμε πολύ καλά το πρόβλημα και τις σχετικέ ε, προκλήσεις. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης κατά νου και αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, με τους εταίρους μας, τις διάφορες οργανώσεις, αλλά και τις οργανώσεις των, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Όχι δηλαδή με μονομένα άτομα, αλλά οργανώσεις οι οποίες πραγματικά διαθέτουν μια τέτοια δομή και κατά συνέπεια έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη ε, και τις δυνατότητες για μια τέτοια συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να αντιταχθούμε στην, στον βιοεξτρεμισμό και την ριζοσπαστικοποίηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να ξεκινήσουμε την συζήτηση να ακούσουμε του βουλευτε Η κυρία χιμενε Μπεσερό. ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διοργάνωση μια τέτοια ακρόαση για ένα τέτοιο θέμα πολύ σημαντικό αλλά και υποτιμημένο σε ό,τι αφορά τη ριζοσπαθικοποίηση στον κόσμο και μια πρωτοβουλία τέτοια η οποία είναι της ε, ομάδας του ΕΛΚ. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν πάρα πολύ χρήσιμε πληροφορίε για το θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο από την Αφρική μέχρι την Ανατολική Ασία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η τρομοκρατία μας πλήττει ενδεχομένως όλους και η ριζοσπαστικοποίηση είναι δραματική παρά την ε, μείωση σε σχέση με τα ποσοστά του 2016. Η ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί μια μεγάλη απειλή ακόμα για την παγκόσμια δημοκρατία. Και έχουμε σχετικές μελέτες στο Μαρόκο, σε hot spot και καταλήγουμε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που προκαλεί ριζοσπαστικοποίηση που αποτρέπει μάλλον την ριζοσπαστικοποίηση είναι οι αξίες και η σχέση με τους φίλους και τον περίγυρο. Αυτό προφανώ έχει ωφέλη για την κοινωνία. Και έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχουν κίνητρα για το άτομο να προβεί σε ριζοσπαστικοποίηση. Είναι λοιπόν κρίσιμο να ελέγξουμε τους παράγοντες αυτούς προκειμένου να μην οδηγήσουν σε ριζοσπαστικοποίηση. Η λύση λοιπόν φαίνεται ότι είναι οι γυναίκες. Η συμπερίληψη λοιπόν των μελών της οικογένειας, των γυναικών της οικογένειας, των αδελφών, των μητέρων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την ε, θεσμική αποτελεσματικότητά μας στην καταπολέμηση ρησπαστικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρείται ότι κατανοεί το ρόλο των ε, γυναικών στην πρόληψη της βίας σε ό,τι αφορά την κατάρτιση μιας στρατηγικής για να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη προς τα θύματα οι παγκόσμιες οργανώσεις κινητοποιούν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να συμμετέχουν πιο πολύ οι γυναίκες και σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες κατά της βίας και της ρεσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα σε φτωχέ χώρες. Για παράδειγμα, ένα ταμείο παγκόσμια ανθεκτικότητα έχει προαγάγει μια πρωτοβουλία κατά την οποία οι γυναίκε θα είναι σημαντικό παράγοντα καταπολέμηση τη βία στην Ιγερία. Το ταμείο αυτό προαγάγει μηνύματα κατά της ριζοσπαθικοποίησης μέσω της συμμετοχής των γυναικών. Και έτσι λοιπόν και στον Παγκλαδές υπάρχουν πρωτοβουλίες τέτοιες για την ε, παροχή αρρωγής προς τις γυναίκες στο Μαλί. Υπάρχει μια, ένα πρόγραμμα κατάρτισης κατά της ριζοσπαστικοποίησης κατά μεγάλο βαθμό συναποτελείται από γυναίκες. Και ο ρόλο των γυναικών σε τέτοιε στρατηγικέ έχει τονιστεί σε διάφορε περιστάσει για τη Συρία, για τον Ιράκ, η ευρωπαϊκή πολιτική, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του 2018 τόνισαν το ρόλο των γυναικών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τέτοιων στοιχείων που οδηγούν τελικά σε ρίζοσπαστικοποίηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, μια προσπαθή μελέτη κατέδειξε ότι 11 ε, μάλλον γυναίκες μέχρι 25 χρονών συγγνώμη, άτομα έως 25 χρονών δήλωσαν ότι όταν αντιμετωπίζουν ένα προσωπικό ή πολιτικό δύσκολο θέμα προτιμούν να στραφούν και να μιλήσουν με τις ε, μητέρες τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στράφηκε λοιπόν στην ε, πτυχή του φίλου σε ό,τι αφορά την αποτροπή της ριζοβαστικοποίησης πρόσφατα. Υπάρχουν παραδείγματα από τις χώρες μέλη, από το ευρωπαϊκό επίπεδο και πρωτοβουλίες κατά πολέμησης της ρίζοσπαθικοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τις εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να κάνω τρία-τέσσερα σύντομα ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Προτιμάτε, Πρόεδρε, να τα θέσω τώρα ή πιο μετά. Πολύ, πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η Πρόεδρος, τώρα, τώρα, αν θέλετε, αλλά σας παρακαλώ πολύ συνοπτικά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό μόνο για τι ερωτήσει σα δίνω. Να σας τα πω στη μητρική μου γλώσσα. Να μου πει παρακαλώ κυρία Μπουζάρ. Πώς αξιολογείται το κατά πόσον λέει ψέματα ή όχι η οικογένεια, η μάνα και γύρω γύρω. Α, γιατί μιλάμε τώρα για τα όσα έγιναν στην ε, Βαρκελώνα. Επί μήνε μήνες οργανωνόντουσαν και κανείς δεν ξέρει τίποτα, ούτε η μάνα, ούτε οι αδερφές, ούτε το παιδί που ήταν ανήλικο, ούτε οι συμμαθητές στο γυμνάσιο, ούτε κανένα. Πώς αξιολογείται λοιπόν το περιβάλλον Επίση. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτός ο πόθος για περιπέτεια, γιατί θέλουν τα παιδιά να είναι κάποιοι που να μην είναι, να μην είναι το, το, το, το, τίποτα. Θέλουν να βγουν από την ανωνυμία, θέλουν να κάνουν κάτι σημαντικό. Τι είπατε? Πώς? Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπέσερα. Συγγνώμη. Sorry, it was her who was telling me to stop. Εσείς μου είπατε να σταματήσω. Εσείς μου είπατε να σταματήσω εκτός μικροφώνου. Okay, okay, I the for that. Νομίζω ότι αυτό είναι δουλειά της Προέδρου. Δεν σα έχω πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Το έχω πει εγώ αυτό. Ποτέ, ποτέ δεν επιτρέπεται. Λυπάμαι, λέει η Πρόεδρο, να συνεχίσουμε και τώρα η κυρία Μπεθέρα. Δύο λεπτά. Το πολύ. Όχι, όχι, ούτε δύο δεν χρειάζομαι. Μα είναι θέμα σεβασμού του άλλου κανείς να χρησιμοποιήσει το χρόνο όσο χρειάζεται. Βέβαια έτσι κι αλλιώς η κατανομή του χρόνου δεν έγινε κατά τέλειο τρόπο ούτε από τις ομιλήτρες. Α, οι ερωτήσεις τώρα. Από πλευράς ευρωπαϊκής, τι γίνεται από πλευράς θεσμικής, από πλευράς προγραμματισμού των πόρων, ούτως ώστε να υπάρχει μια επιχειρησιακή, λειτουργική κάλυψη, γιατί χρειάζεται να δουλέψουμε τι τις ε, γυναίκες παράγοντα της ε, ε, αλλαγής αυτής της μεταξέλιξης δηλαδή έχουμε όλα αυτέ αυτές τις συναντήσεις, τις μελέτες, τις εκθέσεις τι χρειάζεται για να μπορέσουμε στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής οι γυναίκες που είναι το 50% να είναι το, το πρώτο μέσο, το πρώτο εργαλείο, το πρώτο όπλο κατά τη ριζοσπαστικοποίηση. Ευχαριστώ κύριε Νόχιλ. Μία ερώτηση έχω να κάνω και να τη θέσω προ τι εμπειρογνώμονε. Ε, πότε θα πετύχουμε το σημείο σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίηση όπου δεν μιλάμε για ελεύθερη βούληση. Όπου υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο το οποίο έχει ε, πιάσει και έχει φυλακίσει τους ε, νέου. Από ποιο σημείο και μετά δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Πότε δηλαδή είναι ο μαγνήτης τόσο ισχυρό που δεν υπάρχει περιθώριο διαφυγής. Γιατί το θέμα αυτό το συζητάμε και στην ε, υπόθεση της πορνείας. Είναι κάτι άμα ε, εθελούσιο ή πρόκειται για ένα δίχτυ που πιάνει τα άτομα και μετά δεν μπορούν να διαφύγουν. Πού σταματάει δηλαδή η ελεύθερη βούληση και αρχίζει να υπαρχει δρά ο πόλο έλξη τόσο δυναμικά που δεν μπορούν να διαφύγουν πλέον. Αυτό θα με ενδιαφέρει να το ακούσω. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφου, Τη συνάδελφο την Τερέζα που το ε, ξεκίνησε το θέμα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερα επίκαιρο. Άλλωστε αυτά που μα είπαν και οι εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν αυτά που ανέφερε και η Europol προ το Κοινοβούλιο ότι η ριζοσπαστικοποίηση ξεκινά από άτομα που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, σε φυλακές και εκεί πολλοί κόσμος ριζοσπαστικοποιείται. Μεγάλο ποσοστό της ριζοσπαστικοποίησης λαμβάνει χώρα και στο διαδίκτυο και έτσι έγιναν διάφορες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εσείς ε, οι ίδιες ε, διοργανώσατε πολλές τέτοιες έρευνες και φαίνεται ότι τα πορίσματα όλων αυτών των ερευνών δεν καταφτάνουν τελικά στου ε, ηθήνοντε, αυτού που λαμβάνουν τι αποφάσει, για να κατανοήσουν ότι επιτέλου κάτι πρέπει να κάνουμε για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Η κυρία Καρολά. Ανέφερα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Τα ζήσαμε και στο Βέλγιο με τι επιθέσει εδώ. Η ριζοπαστικοποίηση ξεκίνησε από άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ, που έχουν μεγαλώσει εδώ. Και θεωρούσαμε ότι είναι μια χαρά ενσωματωμένα. Δεν είχαν ενσωματωθεί όμω, δεν είχαν ενταχθεί σωστά στην κοινωνία. Ω κοινωνία έχουμε αποτύχει, γιατί αυτά τα άτομα δεν θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σπίτι του, δεν έχουν τι ίδιε αξίε. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτό είναι το ερώτημα. Και ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και του εκπροσώπου ε, τη Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου, οι οποίοι ήρθαν και μα μίλησαν για την κατάσταση στο Βέλγιο. με την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων του Βελγίου σε ό,τι αφορά την αναφορά τους και προκύπτει ότι ο βασικός χώρος ρεζιπαστικοποίησης στο Βέλγιο είναι το κεντρικό τσαμί. Γιατί τα χρήματα προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία. Τα χρήματα τα οποία δεν περνούν από ιονδήποτε έλεγχο. Άρα θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον. Η ριζοσπαστικοποίηση αυτή γίνεται στην Ευρώπη. Και προφανώ θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Ένα άλλο θέμα, ένα άλλο πρόβλημα είναι η κατάσταση στη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Όπου έχουμε όλο και πιο πολλού ε, μαχητέ από τη χώρα αυτή που μεταβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν ότι πολλοί από αυτού του μαχητέ είναι τα γυναίκε. Άρα δεν μεταβαίνουν μόνο εκεί για να βοηθήσουν σε θέματα επιμελητίας. Όχι, έχουν και όπλα. Άρα μου φαίνεται ότι αυτό που διατείνονται πολλοί από τους εμπειρογνώμονες είναι ότι οι αλλοδοποί μαχητές θα πρέπει να ενταχθούν εκ νέου στην κοινωνία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τους ξαναβάλουμε στην Ευρώπη γιατί ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης και αυτό διαφάνηκε από τις σημερινές παρουσιάσεις. Στο θέμα λοιπόν αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον έχετε δεχτεί εσείς επίθεση ή απειλή από Ισλαμιστές σε ριζοσπαστικό παιδικά παράγοντα, γιατί μιλάτε τόσο ανοιχτά για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρεμβάσει σα και λυπάμαι που καθυστέρησα. Δυστυχώ ε, δεν πρόλαβα την παρέμβαση τη κυρία Μπούζο. Να υπενθυμίσω στην κυρία Άιζαξον ότι σήμερα Ο πραγματικός κίνδυνος για τις γυναίκες στην Ευρώπη είναι η Ισλαμική ριζοπαστικοποίηση τα θύματα, οι εκτελέσεις, οι σεξουαλικές επιθέσεις στη Γερμανία. Όλα αυτά τα πρόσφατα περιστατικά καταδεικνύουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της Ισλαμικής ριζοσπαθικοποίησης και είναι εντυπωσιακά λοιπόν τα στοιχεία. Τα θέματα που μας απασχολούν ωστόσο σήμερα. Και εγώ είχα ανταλλαγές απόψεων με πανικολόγους από τη Γαλλία, οι οποίοι μας εξήγησαν πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των γυναικών, ιδιαίτερα στις ευάλωτες περιοχές στη Γαλλία, όπου η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων έχουν κίνδυνο ριζοπαστικοποίησης και προφανώς μετά και κίνδυνο άσκησης τρομοκρατικών επιθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε με τις γυναίκες αυτές, να τις καλέσουμε, να τις ακούσουμε και διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες αυτές φοβούνται. Φοβούνται να βγουν, να μιλήσουν, να καταγγείλουν στην αστυνομία, σε διάφορες οργανώσεις, αυτά που έχουν ζήσει. Και να ακούσουν προφανώς ε, τι έχουμε να τους πούμε. Εσείς τι προτείνετε να κάνουμε. Επίσης, άκουσα να λέτε, κυρία Ζιλ, ότι οι γυναίκες που φορούν ε, μαντήλα υπόκειται στη βούληση του άντρα τους. Σε πολλές περιπτώσεις ακούμε όμως ότι η μαντήλα είναι έκφραση ελευθερία. Είμαστε λοιπόν κάπως προσανατολισμένοι. Τι ακριβώ ισχύει. Και να επανέλθω στο θέμα της οικογένειας, γιατί απασχολεί αυτό και την ε, γαλλική κυβέρνηση. Χθες προχθές ακούσαμε ότι πολλά παιδιά στο σχολείο αρνούνται όλο και πιο πολύ να κάνουν παρέα με παιδιά τα οποία δεν είναι μουσουλμανοί. Αυτό από μία έρευνα λοιπόν της ε, γαλλικής ε, κυβέρνησης και δεν θέλουν να ακούν τη μουσική, δεν θέλουν τα αγοράκια να κρατάνε τα χέρια από τα κοριτσάκια. Αρνούνται ακόμα να κάτσουν και δίπλα σε κάποιον ο οποίος δεν τρώει χαλάλ ή τρώει α, Πώ μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε αυτέ τι οικογένειε. και πώ μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, προτού πάνε στο σχολείο. Ευχαριστώ και τώρα το λέγουν και πάλι οι εμπειρογνώμονε μα για να ακούσουμε σχόλια, απαντήσει, παρατηρήσει. Παρακαλώ να θυμάστε ότι έχετε δύο λεπτά η κάθε μία, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ και πια θα ξεκινήσει. Ε, je, je avec vous, que... Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, για να μην την ξεχάσω. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τη μαντήλα δεν με καταλάβατε. Αυτό που είπα είναι ότι είναι στερεότυπο το οποίο επικρατεί. Είναι η ευθύνη της γυναίκας τζιχαντίστριας ενδεχομένω. Και αυτό μπορεί να προκύψει από μια επέκταση του ρατσισμού που επικρατεί στην Γαλλία αυτό το στερεότυπο που υπάρχει ότι μία ε, γυναίκα μουσουλμάνα δεν είναι ελεύθερη γιατί δεν ε, μπορεί να ασκήσει τις επιλογές της. Δεν είχε να κάνει με τη μαντήλα αυτό που είπα. Και πιστεύω ότι η άγνοια αυτή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μας ε, οδηγούν στο να κάνουμε λάθος και να μην αξιολογούμε σωστά την κατάσταση αυτή, δηλαδή η έλλειψη δίθεν αυτό διάθεση των γυναικών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτά κατά περίπτωση για να εμβαθύνουμε λίγο τη συζήτηση και θέλω να κατανοήσω ότι η γυναίκα είτε είναι ε, υπεύθυνη είτε όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τις γυναίκες. Ε, πιστεύω ότι έχουν μεγάλο ρόλο να δραματίσουν τα μέσα ενημέρωση και θα πρέπει οι μητέρε οι γυναίκες να παρουσιάσουν και να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους, τις ιστορίες τους σε μικρές ε, επιτροπές ε, όταν τους δίνουμε την ευκαιρία. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία αναφέρω στο βιβλίο μου, η οποία προσπαθεί να στραφεί σε σχολεία, σε μικρές κοινότητες και να αναφέρει τι έζησε, τις μαρτυρίες της σε σχέση με το γιο της. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι μαζί να καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου να κατανοήσουμε τον εχθρό και να κατανοήσουν και οι γυναίκες ότι έχουν φωνή. Έχουν φωνή και έχουν και ευθύνη έναντι της κοινωνίας. Γιατί αυτές που έχουν πληχτεί από το φαινόμενο έχουν να πούν πιο πολλά σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόληψης. Ευχαριστώ. Εγώ θα δώσω το λεπτό που μου αναλογεί στην κυρία Ιζαξόν και στην κυρία Γκαρσία για να αντισταθμίσουμε λίγο την ανισότητα που ήταν επικράτησε στην αρχή, στον χρόνο παρέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, να πω όμω και ότι και οι τέσσερι μιλήσαμε για τι ταξικέ διαφορέ, για για τις οικογένειες που έχουν πληχθεί από τη ριζοσπαστικοποίηση. Και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε διαδικασία, χρόνο να μιλήσουμε για τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίηση και οι τέσσερις είπαμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, ποιε τάξει πλήττονται πιο πολύ. και θεωρείται πάντα ότι πρόκειται για πεθοεμπρεμένου ε, μουσουλμάνους ε, που δεν έχουν ευκαιρίε στη ζωή. Αυτό από επιστημονική άποψη δεν στέκει. Αν μείνει σε τέτοιο συναισθηματικό επίπεδο η συζήτηση να προστατεύσουμε τον κόσμο γιατί φταίνε αυτοί οι ή οι μουσουλμάνοι και το καθεξής, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Δεν θα κουνήσουμε ρούπι και σα δίνω το λόγο παρά αυτά. Για να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε η κυρία Μπεθέρα. Με δύο πινελιέ έχουν να πω ότι δεν θα πρέπει κανεί να υιοθετεί θέσει ελιτίστικε. Θα προσπαθεί κανεί να έχει μία ε, έποψη από κάτω προ τα πάνω, από τη βάση ε, και οριζόντια. Ε, ε, έτσι, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν πολύ καλά την ουσία και τη βάση. Ε, ούτως είπε, ε, γιατί είπαμε ποιες είναι όλες οικογένειας των γυναικών, αυτών που βοηθούν στο σπίτι, είναι, είναι επαγγελματίε. είναι κάποιοι ειδικοί που τα ξέρουν και μπορούν να βοηθήσουν τη λήψη των αποφάσεων. Κάτι άλλο επίσημα σημαντικό είναι το ότι θα πρέπει να απο γυμνωθεί να ξεκαθαριστεί από γυναίκες αυτός ο κλάδος γιατί αυτό πολλές φορές το κάνουν τα κράτη ε, και αυτό το οποίο χρειάζεται όμως είναι να βελτιωθεί το ότι όλο ένα και περισσότερες γυναίκες ε, συμμετέχουν μα μια που δεν έχουμε χρόνο να σας πω μόνο μόνο μόνο με λίγα λόγια ε, τι γίνεται με αυτό το δίπολο σχετικό με την ένταξη, γιατί λέμε για την ένταξη κάπως απλουστευτικά από πλευράς κοινωνικονομικής ή από πλευράς πολιτιστικής πρόκειται για κάποιο σωστικοποίηση που γίνεται βία. Μα γίνεται, ναι, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά προφίλ, οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλούμε περισσότερο για τελικά έλλειψη αφομοίωσης πολιτιστικής Πολλές φορές έχουμε κάποιες που έχουν δουλειά, ξέρουν τη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά όμως πολιτιστικά δεν αφομοιώνονται. Το είδαμε και στην Ισπανία, είναι πάρα πολλές. Ε, πολλοί αυτοί νέοι που έρχονται. Ε, στην Ισπανία έρχονται από το Μαρόκο, ναι, πολλές φορές όμως ε, ε, ε, υπάρχουν και κάποιοι Ευρωπαίοι. Ε, ασυμμετρία, είναι θέμα παιδείας επίσης. Να, και στο Ριπόλ και στο Καμπρίλς έτσι λειτουργήσε ε, εκείνη η τρομοκρατική ομάδα. Και όσον αφορά τις γυναίκες στην Ισπανία δεν υπήρχε προηγούμενο, δεν είχαν ποινικό μητρό, τίποτα, τίποτα. Ούτε πτέσμα δεν είχαν κάνει και ε, είπαμε ότι αυτό καμιά φορά συντρέχει για, τις, τους αλλά όχι για τις γυναίκες. Ε, είναι φιλοσοφικό το θέμα αυτό, ενδεχομένω το τι είναι θελούσιο και τι όχι, πού σταματάει η ελεύθερη βούληση. Είμαι εδώ γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Ε, εν πάση περιπτώσει. Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξετήσουμε όταν μιλάμε για τον εθελούσιο χαρακτήρα είναι το πλαίσιο. Ποια είναι η δηλαδή, τι εναλλακτική υπάρχει. σε ό,τι αφορά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους. Και φυσικά σε ό,τι αφορά την ε, πορνεία που αναφέρατε, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για την βίαιη πορνογραφία. Δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό για τη δική σας ερώτηση. Δεν είδα το όνομά σας να σας πω απλά ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ας το αφήσουμε εκεί. Υπάρχουν διάφορες τύποι ριζοπαστικοποίησης και βίαιης, βίαιου εξτρεμισμού. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδεχομένως πολιτική σκοπιμότητα για την πρόθεση της βίας. Εμάς δική μας δουλειά είναι να είμαστε αντικειμενικοί. Μιλάμε με εκπροσώπους ε, του Σώματος Επιβολής του Νόμου, των δικαστών, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τι είναι επικίνδυνο και βίο για τη γυναίκα και εδώ στην Επιτροπή σας τα γνωρίζετε αυτά ότι αυτό δεν είναι τίποτα σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη ριζοπαθικοποίηση. Το πρόβλημα, ξέρετε ότι είναι πιο μεγάλο όταν πρόκειται για τον σύντροφο ζωής, τον σύζυγο μέσα στο σπίτι των γυναικών. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία για το ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο για μια γυναίκα. Νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρα κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ του εμπειρογνώμονε. τι εμπειρογνώμονε, μάλλον, λέει η Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ και εσά και του βουλευτέ για την ενεργό συμμετοχή στην ακρόαση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ.